Συνάδελφοι, καλησπέρα. Εγκρίνεται η μερίσια διάταξη αν δεν έχετε παρατηρήσεις. Δεν υπάρχουν σχόλια από τον Πρόεδρο, ανακοινώσεις. Ε, κροατικά, δανέζικα, λετωνικά, αγγέλικ δεν θα έχουμε στη διερμηνία σήμερα. Είναι πιο σύντομη η συνεδρίασή μας από ό,τι συνήθως και περνάμε ευθύ αμέσως στο πρώτο σημείο στην ημερήσια διάταξη που σήμερα γενικά η συνεδρίασή μας είναι αφιερωμένη στη μετανάστευση. Το πρώτο θέμα λοιπόν είναι ανταλλαγή απόψεων ε, για τη συνέχεια που δόθηκε στη διακήρυξη της Νέας Υόρκης με παρουσίαση της Έλεν Χάντσεν που είναι κύριε Σύμβουλος Πολιτικής της ΥΠΑ της Αρμοστίας των ΗΠΑ Εθνών για τους πρόσφυγες σχετικά με το Παγκόσμιο Σύμφωνο για το προσφυγικό και τον Μαμάντου Μπέιλ, που είναι πληρωτή διευθυντή τη ομάδα CRRF, e το πλαίσιο ολοκληρωμένη απάντηση στο ζήτημα των προσφύγων. Θα θυμόσαστε ότι τη 19 Σεπτεμβρίου αποφασίσαμε να αντιμετωπίσουμε κάποια στιγμή, να συζητήσουμε αυτό το μεγάλο θέμα των προσφύγων και των μεταναστών. Και θα θυμόσαστε ότι μετά από την ε, διάσκεψη που έγινε τότε αποφασίστηκε να δοθεί καλύτερη απάντηση στις προκλήσεις αυτές και η απάντηση αυτή είναι αυτό που ονομάζουμε διακήρυξη της Νέας Υόρκης. Θα θυμόσαστε τη συζήτηση που είχαμε κάνει τότε. Το Κοινοβούλιο ήταν παρόν βέβαια σε αυτήν την ε, διάσκεψη. Είχαμε τρία μέλη, την κυρία Βίλστρομ, την κυρία Σφάιν από την Επιτροπή μας και συμμετείχε η αντιπροσωπεία αυτή επίσης και σε μια συνάντηση τον Ιανουάριο. Έτσι λοιπόν προσκαλέσαμε την Αρμοστία να έρθει στην Επιτροπή μας να συζητήσει μαζί μας αυτά τα τόσο σημαντικά θέματα. Και συμφωνήσαμε επίσης να κάνουμε και μια χωριστή συζήτηση για το σύμφωνο όσον αφορά τους μετανάστες. Έχει δοθεί ιδιαίτερη σημασία στο θέμα και από εμά και από την Αναπτυξιακή Επιτροπή και από την Επιτροπή Εξωτερικών Υποθέσεων του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Και μετά το καλοκαίρι θα έχουμε και μια δεύτερη ανταλλαγή απόψεων με συγκεκριμένες χώρες. Ελπίζω επίσης να έρθει και ο κ. Δεγκράντη που είναι ο ύπατος αρμοστής για το θέμα, το μεταναστευτικό. Έτσι καλώ στην Ολομέλεια θα έρθει ο Γενικός Γραμματέας του ΟΗΕ και θα μιλήσει σε εμά για το μεταναστευτικό και το προσφυγικό. Στα πλαίσια αυτά λοιπόν νομίζω ότι ήρθε η ώρα να ακούσουμε τους προσκεκλημένους μας. Θα ακούσουμε πρώτα απ' όλα την κυρία Έλεν Χάνσεν που είναι κύρια σύμβουλος, όπως είπαμε, πολιτικής της ΥΠΑ Αρμοστίας και θα μας μιλήσει για το σύμφωνο αυτό, το παγκόσμιο για τους πρόσφυγες. 10-15 λεπτά παρακαλώ. Παρακαλώ κύριε Χάνισεν, έχετε το λόγο. Ε, Ξιότιμε Πρόεδρε, κυρίες και κύριοι, ευχαριστώ πολύ στην είπατε αρμοστία εκτιμούμε όλος ιδιαίτερος το ενδιαφέρον που δείχνετε αλλά και τη δέσμευση που έχετε, αναλάβετε, που έχετε αναλάβει, συγγνώμη, όπως επίσης και την καλή συνεργασία που έχουμε μεταξύ μας μέχρι τώρα. Θέλω να πάμε λίγο πριν τη 19η Σεπτεμβρίου, τότε δηλαδή που εγκρίθηκε η διακήρυξη. Ποιο ήταν το πλαίσιο τότε. Είχαμε πάνω από ένα εκατομμύριο που φτάνανε στην ε, Ευρώπη το 2015, μην ξεχνάμε, και η κατάσταση ήταν χωρίς προηγούμενο όσον αφορά τη μετατόπιση πληθυσμού ανά το κόσμο. Η διεθνή κοινότητα όμως τελικά είπε κάτι πρέπει να κάνουμε και με την όθηση του ΟΙΕ. Φιλοξενούν ε, πρόσφυγες πολλές χώρες του κόσμου και θα εξακολουθούν για μεγάλο χρονικό διάστημα. Ο κύριος ε, Μπάλτη θα μιλήσει περισσότερο για αυτό το ζήτημα σε λίγο. Πάντως όσον αφορά την ε, διάσκεψη της Νέας Υόρκης, περιλαμβάνει δεσμεύσεις από τις χώρες μέλη υπέρ των προσφύγων και των μεταναστών. Είναι μια δέσμευση από κοινού που αναλαμβάνουμε και υπάρχουν και ειδικέ δεσμεύσεις. Από τη μια μεριά για τους μετανάστες για μια διαδικασία η οποία θα ακολουθήσει σε ένα παγκόσμιο σύμφωνο υπέρ μιας ασφαλούς μετανάστευσης που θέλουμε να εγκριθεί το 2018. Η διαδικασία αυτή πάντως είναι μια διαδικασία της οποίας ηγήθηκαν οι χώρες μέλη και διευκολύνθηκε και από την Ελβετία και το Μεξικό τους αντιπροσώπους των χωρών αυτών στον ΟΗΕ δηλαδή στη Νέα Υόρκη. Το πρώτο παράστημα λέει ποια είναι η απάντηση και ζητάει από τον Νόιε να εκπονήσει πλαίσιο για ανταπόκριση στο προσφυγικό προστατεύοντας μεγάλα τμήματα του πληθυσμού. Ο κύριος Ζουμπάλτη είναι αυτός που θα αναφερθεί περισσότερο στο, στην ανταπόκριση αυτή. Πάντως αυτή η ανταπόκριση αφού αξιολογηθεί θα οδηγήσει τελικά στο Παγκόσμιο Σύμφωνο για τους πρόσφυγες το οποίο θα βασίζεται κύρια στην ανταπόκριση αυτή που θα ετοιμάσουμε για το προσφυγικό. Ο ύπατος ε, αρμοστής θα το συμπεριλάβει στην ετήσια εκθεσή του προς τον Γενικό Γραμματέα το 2018 και η έκθεση αυτή θα τελειώσει τον Ιούλιο-Αύγουστο του 2018 και θα περιλαμβάνει και το Παγκόσμιο Αυτό Σύμφωνο. Στη συνέχεια θα πάει στην Γενική Συνέλευση του ΟΓΕ το 2018 και θα εγκριθεί μαζί με το ψήφισμα της Γενικής Συνέλευσης όσον αφορά το έργο της ύπατης αρμοστίας του ΟΗΕ για τους πρόσφυγες. Αυτό κανονικά θα γίνει τον Νοέμβριο του 2018. Τώρα για να επανέλθουμε όμως λίγο στο τι θα προηγηθεί του, της Γενικής Συνέλευσης. Όπως σας είπα, ηγούνται τα κράτη-μέλη και βοηθούν πολύ οι βόρειες χώρες. Η Σουηδία αυτή τη φορά, το 2018, θα διευκολύνει τη διαδικασία έγκρισης του ψηφίσματος που θα περιλαμβάνει κανονικά μία παράγραφο που θα λέει ότι εγκρίνεται το Παγκόσμιο Σύμφωνο. Λοιπόν, για να επανέλθουμε λίγο στο τι θα είναι αυτό το Παγκόσμιο Σύμφωνο. Είπα ότι η Ερμοστή για τους πρόσφυγες έχει ετοιμάσει ένα χάρτη πορείας για το σύμφωνο αυτό, το οποίο το γνωρίζετε. Αν δεν το γνωρίζετε, να ξέρετε είναι στην ιστοσελίδα μας. Στην αρχική σελίδα. Και ο τρόπος που εμείς το αντιμετωπίζουμε είναι ότι θα είναι η απα... το πλαίσιο απάντησής μας στο προσφυγικό έτσι όπως έχει στη διακήρυξη της Νέας Υόρκης, χωρίς να το πειράξουμε, θα υπάρξουν κάποια προήμια που θα λένε ότι επιβεβαιώνουμε τις δεσμεύσεις ε, όσον αφορά την προστασία ε, των προσφύγων κτλ. Και θα υπάρχουν και κάποιες παράγραφοι στο τέλος οι οποίες θα λένε ποιο θα είναι το δεύτερο μέρος του Παγκοσμίου Συμφώνου. Το δεύτερο τμήμα του Παγκοσμίου Συμφώνου θα είναι το πρόγραμμα δράσης. Πρόγραμμα δράσεις που θα περιλαμβάνει στοιχεία τα οποία θα περνούν στην εφαρμογή των δεσμεύσεων που έχουν λάβει οι χώρες μέλη του ΟΗΕ στην ε, δήλωση που θα αναφέρεται στο ψηφίσμα με την απάντησή μας στο προσφυγικό. Δύο τμήματα λοιπόν. Το ένα είναι το πλαίσιο για την απάντηση στο προσφυγικό και το δεύτερο είναι το πρόγραμμα δράσης. Προκειμένου τώρα να καταλήξουμε στο πρόγραμμα δράσης, έχουμε συναντήσεις, διαβουλεύσεις, πρώτα απ' όλα ετήσιες διαβουλεύσεις με τις μη κυβερνητικέ οργανώσεις ήδη φέτος. Στο δεύτερο εξάμεινο της χρονιάς αυτής θα οργανώσουμε και κάποιες θεματικές συναντήσεις. Εκεί θα ακολουθήσουμε βέβαια την συνολική μας απάντηση στο προσφυγικό. Θα αναφερθεί σε αυτό περισσότερο ο κύριος Μπάλτη. Και μετά θα δούμε και ποια είναι η κατάσταση, δηλαδή πώς το πλαίσιο αυτό απάντησης συνολικά στο προσφυγικό, πώς θα μας προσφέρει την αλλαγή αυτή που χρειαζόμαστε στον τρόπο με τον οποίο λειτουργούμε και μετά θα υπάρχει ο διάλογος 12 και 13 Σεπτεμβρίου με τον ύπατο αρμοστή για το προσφυγικό. Συζήτηση δηλαδή μεταξύ χωρών μελών, εμπειρογνωμόνων, μη κυβερνητικών οργανώσεων, άλλων ε, οργανώσεων και τον Φεβρουάριο του 2019 ο Ήπατος αρμοστής θα προτείνει και ένα αντίγραφο του συμφώνου αυτού. Και μετά θα αρχίσουν επίσημα διαβουλεύσεις με τις χώρες μέλη του ΟΗΕ. Ακόμα όμως βέβαια που είναι πολύ ιδιαίτερη η διακήρυξη της Νέας Υόρκης για τον Υπατορμοστή, ότι δηλαδή μπορεί να βάλει στην ετήσια εκθεσή του προς τη Γενική Συνέλευση ο Ήπατος στην αξιολόγησή μας και αυτό είπαμε ότι θα το κάνουμε μετά από διαβούλευση με τους εταίρους μας. Χρειάζεται οπωσδήποτε να έχουμε ένα κείμενο πάνω στο οποίο να υπάρξει ευρεία συνένεση ώστε να εγκριθεί από την Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ στα τέλη του 2018. Γι' αυτό λοιπόν ξεκινούμε πρώτα με άτυπες διαβουλεύσεις, με καταγραφή της κατάστασης και μετά με επίσημες διαβουλεύσεις. Το πρώτο εξάμενο της επόμενης χρονιάς. Όλα αυτά αναφέρονται στο χάρτη πορείας μας. Θα επανέλθω μάλλον προηγουμένως να πω κάτι ακόμα. Ότι αυτό που μας ενδιαφέρει είναι η ασφάλεια των προσφύγων και των μεταναστών και γι' αυτό προβλέπουμε δύο διαφορετικές και ανεξάρτητες μεταξύ τους διαδικασίες. Θα υπάρχουν δύο διαφορετικές διαδικασίες λοιπόν, αλλά θα συνεργαστούμε με τους εταίρους μας ώστε να υπάρχει συμπληρωματικότητα μεταξύ των δύο συμφώνων και να υπάρχουν κοινέ δεσμεύσει που να ακολουθούν και τις δύο διαδικασίες. Για παράδειγμα, η λαθροδιακίνηση, η διάσωση στη θάλασσα, η αντιμετώπιση ειδικών αναγκών. Όλα αυτά λαμβάνονται υπόψη και στις δύο περιπτώσεις. Είτε πρόκειται δηλαδή για τους πρόσφυγες, είτε πρόκειται για τους μετανάστες. Αυτά θα είναι τα δύο σύμφωνα. Τώρα, έρχομαι ειδικότερα στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Κοίταζα το Lives and Dignity, που είναι η πολιτική του 2016 και πρέπει να σας πω ότι εκπλήσεται κανείς από τη συμπληρωματικότητα και την συνέπεια των ε, πολιτικών στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Και θυμίζουν πολύ τη συνολική αυτή απάντηση του ΟΙΕ. Ε, χρησιμοποιείται η ίδια γλώσσα για να αντιμετωπιστούν οι ρίζες του προβλήματος, υπογραμμίζεται το θέμα της συμμετοχής όλων υπογραμμίζεται η ανθρωπιστική αρρωγή, η συνεργασία προς την επίτευξη κοινών στόχων, ε, να προχωρούμε βάσει στοιχείων και δεδομένων, το να βρίσκουμε έγκαιρα λύσεις. Με δύο λόγια πιστεύουμε ότι είμαστε απόλυτα συμπληρωματικοί μεταξύ μας. Συνεπώς το πρώτο μήνυμα που θέλω εδώ να περάσω είναι αυτό. Η συμπληρωματικότητα και η συνέπεια των πολιτικών της Ευρωπαϊκής Ένωσης μαζί με αυτά που εμείς προσπαθούμε να πετύχουμε στον ΟΗΕ. Και έτσι, για μας η Ευρώπη είναι ο πρωταθλητής της συνολικής αυτής απάντησης στο προσφυγικό. Πάντως η διακήρυξη της Νέας Υόρκης προσφέρει κατευθυντήριες γραμμές προς πάσα κατεύθυνση για το πώς να προχωρήσουμε. Άρα και για την Ευρώπη. Μερικές φορές ο κόσμος νομίζει ότι ο ρόλος της Ευρώπης είναι χρηματοδότηση ώστε να κρατήσει τους μετανάστες και τους πρόσφυγες μακριά από τα σύνορά της. Εμείς πιστεύουμε ότι υπάρχουν και κάποια καλά στοιχεία για τα πρόπτα, για την συμμετοχή όλων, Τέλος, νομίζω ότι πολλά μπορούμε να πούμε για το μήνυμα που πρέπει να περνάμε στον κόσμο για αυτό που έχουμε ακούσει ως κρίση, προσφυγική κρίση, μεταναστευτική κρίση. Όμως στην πραγματικότητα εμείς πιστεύουμε ότι αν γίνονται ε, σημαντικές προσπάθειες ώστε να προχωρούμε χέρι-χέρι με διεθνή συνεργασία και μοιραστούμε πραγματικά τις ευθύνε και τις αρμοδιότητες, τέτοιες καταστάσεις είναι διαχειρίσιμες. Αλλά χρειάζονται μια πραγματική εταιρική σχέση, πραγματική συνεργασία. Όσον αφορά την Ευρώπη, εμείς θέλουμε να υπάρχει συμπληρωματικότητα πόρων και στην ανθρωπιστική βοήθεια. Θέλουμε επιπλέον βοήθεια όσον αφορά τη συνολική μας απάντηση στο προσφυγικό ένας τομέας σχετικά με τον οποίο πιστεύουμε ότι οι ευρωπαϊκές χώρες μέλη θα μπορούσαν να κάνουν παραπάνω προσπάθεια είναι στο θέμα της επανεκατάστασης και των νόμιμων διόδων μετανάστευση. Έχω πάει και στην Ελλάδα και μίλησα εκεί με μία 80χρονη η οποία είχε πάρει το πλοίο γιατί ήταν ο μόνος τρόπος για να ξαναβρει την οικογένειά της σε ευρωπαϊκές χώρες μέλη. Η επανεγκατάσταση λοιπόν και άλλες ασφαλή δίωδοι είναι ό,τι καλύτερο έχουμε να προσφέρουμε. Και εφόσον εφαρμοστεί αυτό, στέλνουμε και ένα πολύ καλό μήνυμα στις χώρες που φιλοξενούν πρόσφυγες. Για το 86% των προσφύγων βρίσκονται σε νότιο ημισφαίριο, σε φτωχές χώρες, και όχι στη, στον πλούσιο βορρά. Αυτό λοιπόν είναι πολύ σημαντικό, να στείλουμε δηλαδή αυτό το μήνυμα ότι μοιραζόμαστε τις ευθύνες. Γιατί έτσι με απτές αποδείξεις ότι μοιραζόμαστε την ευθύνη, μπορούμε να προχωρήσουμε. Αν δεν υπάρχει αυτή η απτή απόδειξη για αυτές τις φτωχές χώρες, δύσκολα θα μπορέσουν να αντέξουν το βάρος και τον αντίκτυπο αυτών των τεράστιων ροών που έχουν καταλήξει στις χώρες αυτές. Αυτά, Πρόεδρε, και τώρα μου επιτρέπετε να δώσω το λόγο στον κύριο Μπάλτη για τη συνέχεια. Ευχαριστώ. Σας ευχαριστώ. Αξιότιμη κύριε Πρόεδρε, κυρίες και κύριοι, εγώ θα ήθελα να συμπληρώσω τα όσα είπε η κυρία Χάνσεν μόλις, τονίζοντας τρία ζητήματα. Το ένα είναι ότι θα πρέπει να θυμηθούμε τον στόχο του συνολικού πλαισίου ανταπόκρισης στους πρόσφυγες που βρισκόμαστε αυτή τη στιγμή γιατί αυτή είναι μια έκκληση που έχουν κάνει τα κράτη ε, της Ευρωπαϊκής Ένωσης προς την UNHCR, την είπατε αρμοστία για τους πρόσφυγες του ΟΗΕ Ο λόγος ύπαρξης αυτού του πλαισίου για τους πρόσφυγες είναι πρώτον να διευκολυνθεί, να αυλυνθεί η πίεση στις χώρες ε, που φιλοξενούν τεράστιους αριθμούς προσφύγων που κάποιες φορές ανέρχονται μάλιστα στο 10% ε, σε σχέση με το πληθυσμό κάποιας χώρας και έχουμε δει πολλές από αυτές τις χώρες. Το δεύτερο αφορά την ε, αύξηση της ανεξαρτησίας των ε, προσφύγων μέχρι ότου με αξιοπρεπή τρόπο να μπορέσουν να βρουν πιο μόνιμες λύσεις και έπειτα να δούμε ποιες λύσεις τρίτων χωρών μπορούν να υπάρξουν μέσω της επανεγκατάστασης σε μεγάλους βαθμού, αριθμούς αλλά ξέρουμε ότι η επανεγκατάσταση δεν είναι απαραίτητο η μόνη απάντηση αν και γνωρίζουμε πως συμβάλλει στην ε, μείωση ε, των προβλημάτων και διευκολύνει αλλά εκτός από την επανεγκατάσταση κάνουμε ε, ε, γενιακή επανένωση καθώς και επιπλέον στήριξη μέσω, για παράδειγμα, της ε, μετανάστευσης για λόγους εργασίας. Τέταρτο στοιχείο είναι η δημιουργία των προϋποθέσεων στις χώρες προέλευσης ώστε οι ε, πρόσφυγες να μπορούν ενήμεροι πλέον να επαστρέψουν εθελοντικά στις χώρες τους, να μπορούν να βρουν δηλαδή λύσεις μόνιμες μέσω στηριζόμενης εθελοντικής επιστροφής. Αυτά προβλέπει το καθολικό πλαίσιο για τους πρόσφυγες, ε, αυτά που συμφωνήθηκαν στη διακήρυξη της Νέας Υόρκης το 2016. Think... θέλω να σας πω που βρισκόμαστε μια μέρα μετά τη δήλωση της Νέας Υόρκης ε, της 19 Σεπτεμβρίου πολλές χώρες ανέλαβαν δεσμεύσεις, ε, έκαναν υποσχέσεις και μέχρι σήμερα μπορούμε να πούμε ότι υπάρχουν κάποιες χώρες, ιδιαίτερα στην Αφρική, που έχουν δεχτεί να χρησιμοποιηθούν ως χώρες πιλωτικές για την υλοποίηση αυτού του προγράμματος. Πρώτα είναι η Ουγγάντα, νομίζω που μόνο με 35 εκατομμύρια πληθυσμό έχει δεχτεί πάνω από ένα εκατομμύριο πρόσφυγες. Ε, ε, δείχνει αυτό τη γενεοδορία της χώρας αυτής απέναντι στους γείτονες από τον Νότιο Σουδάν, την Σομαλία και κάποιες ακόμα χώρα. Επιπλέον από τη Ουγγάντα που ακόμα αντιμετωπίζει επίγουσες ανάγκες αλλά και παρατεταμέν, φιλοξενεί παρατεταμένες ε, προσφυγικούς πληθυσμούς. Έχουμε την Τανζανία που έχει ανοίξει τις πύλες της σε εκατοντάδες χιλιάδες πρόσφυγες στις τελευταίες δεκαετίες και επίσης έχει χρησιμοποιηθεί ως χώρα ε, ε, πιλωτική. Μετά έχουμε την Αιθιοπία και το Τζιμπουτί. Η Αιθιοπία και το Τζιμπουτί και εδώ θα σταθώ σε αυτές τις χώρες για λίγα λεπτά, γιατί αυτές οι χώρες παρά τη γενοδορία τους λάμβαναν και δέχονταν μεγάλους αριθμούς προσφύγων, αλλά δεν άνοιγαν απαραίτητο στην αγορά εργασίας τους. Χάρη στις υποσχέσεις που ανέλαβαν στις 20 Σεπτεμβρίου πέρυσι, Υπήρξε μια μετακίνηση της πολιτικής ώστε να εξασφαλιστεί ότι το Τζιμπουτί αλλά και η Αιθιοπία θα συνεχίσουν να βοηθούν ε, πρόσφυγες να ζουν μια αξιοπρεπή ζωή. Και η Σομαλία είναι σημείο εστίασης. Και ξέρουμε πως η Ευρωπαϊκή Ένωση έκανε μια διάσκεψη κορυφής για τους πρόσφυγες που αφορούσε το άσυλο αλλά και τη δημιουργία προϋποθέσεων ώστε να βοηθηθούν οι πρόσφυγες που επιθυμούν να επιστρέψουν στις χώρες τους. Πέρα από την Αφρική είδαμε κάποια ενδιαφέροντα στοιχεία σε σχέση με τη Γουατεμάλα, όπου συνεχίζεται η συζήτηση για να δούμε αν επιπλέον χώρες θα δεχτούν να χρησιμοποιηθούν ως χώρες εστίασης για το ε, καθολικό σύμφωνο για τους πρόσφυγες. Αυτό που επίσης βλέπουμε είναι ότι δεν θα πρέπει να εστιάσουμε μόνο στις χώρες που προσπαθούν να δείξουν προθυμία ώστε να χρησιμοποιηθούν ως χώρες CRRF, δηλαδή του Συμφώνου για τους πρόσφυγες. Αλλά όπως είπε και η συνάδελφος Χάνσεν προηγουμένως, θέλουμε και προσβλέπουμε στην Ένωση να συνεχίσει να βοηθάει και να στηρίζει χώρες που αποτελούν ε, σημεία εστιασμού για το σύμφωνο για τους πρόσφυγες και που δέχονται το μεγαλύτερο μέρος των προσφύγων παγκοσμίως ε, αλλά και που ξεπερνούν και τους εαυτούς τους, γιατί υπάρχουν και πολλές άλλες χώρες που δεν δέχονται να γίνουν ε, χώρες εστιασμού. Κάτι ακόμα που είναι πολύ σημαντικό είναι να δούμε ότι αυτό το σύμφωνο για τους ε, πρόσφυγες ε, που είναι ένα μέσο μοιρασιά, ας πούμε, των προσφύγων, δίκαιες μοιρασιάς των προσφύγων, να μην χρησιμοποιηθεί ως μέσο ώστε να μείνουν μονίμως κάπου σε συγκεκριμένε χώρε οι πρόσφυγες Να αυξηθούν οι δυνατότητε για επανένωση οικογενειών, για επανεγκατάσταση και επίσης αυτό τώρα είναι το τελευταίο κομμάτι της παρέμβασής μου ότι θα πρέπει να επικρατήσει μια προσέγγιση από πλευρά ολόκληρη τη κοινωνία. Εμεί, οι κυβερνήσει, οι εκπρόσωποι των κυβερνήσεων, τα εκτελεστικά σώματα, τα δικαστικά σώματα, θα πρέπει να ε, τίνουμε χείρα προ την κοινωνία των πολιτών αλλά και προ του ίδιου του πρόσφυγε Αυτό νομίζω ε, θα πρέπει να γίνει. Γενική συνεργασία. Ευχαριστώ πολύ. Ε, οι συνάδελφοι θέλουν να καταλάβουν ακριβώς τι σημαίνει αυτό το Global Compact, το σύμφωνο, στην πράξη. Πριν τους δώσω το λόγο, ήθελα στην αρχή να δώσω ένα είδος χρονοδιάγραμμα για το πώς θα συνεχίσουμε να συμμετέχουμε στην διαδικασία του Global Compact του Παγκόσμιου Αυτού Συμφώνου. Στο τέλος θα έχουμε κάποιες παρεμβάσεις μεταξύ αυτών και μία σχετικά με τη συμμετοχή μας στον διάλογο του είπα Ελπίζω σε συνεργασία με την Υπηρεσία Εξωτερικών Δράσεων τον Δεκέμβριο. Ας ακούσουμε τώρα την σύντομη παρέμβαση της Υπηρεσίας Εξωτερικών Δράσεων. Έχετε το λόγο. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε που μας δίνετε την ευκαιρία να δώσουμε ένα σύντομο, μια σύντομη σκιαγράφηση τη συμμετοχή της Ευρωπαϊκή Ένωση στη διαδικασία για την σύνταξη των δύο, ε, συμφωνιών. Είναι σαφές ότι χρειαζόμαστε μια συνολική προσέγγιση αν θέλουμε να απαντήσουμε στις προκλήσεις ε, της ε, αναγκαστικής μετακίνησης. Όπως ελέγχθηκε πριν, η Ευρωπαϊκή Ένωση είναι πρωτοπόρος στην αυτή προσέγγιση με την ανακοίνωσή μας Life and Dignity του Απριλίου του 2016 που αναζητήσαμε μια συνολική προσέγγιση για τις αναγκαστικές μετακινήσεις. Ως αποτέλεσμα, η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει αυξήσει σημαντικά τις προσπάθειες για να αντιμετωπίσει την αναγκαστική μετακίνηση ιδίως στην Ανατολική Αφρική και στην Ασία. Η εργασία αυτή είναι συμπληρωματική με τη διαδικασία RRF και κινείται στην ίδια κατεύθυνση. Και καλωσορίζουμε πολύ τη διαδικασία αυτή γιατί είναι και μια ευκαιρία για μας να δώσουμε εντονότερη ορατότητα στις δικές μας πρωτοβουλίες που έχουν σχέση με την προστασία και στη συνεργασία με τρίτες χώρες. Θεωρούμε ότι το CRRF είναι καλή βάση για την ανάπτυξη ενός Global Compact υπέρ των προσφύγων και χαιρόμαστε για τον κεντρικό ρόλο που παίζει ο υπάτος αρμοστής. Η Ευρωπαϊκή Ένωση mm. αναμειγνύεται στη διαδικασία από τα πρώιμα στάδια με τις αντιπροσωπείς μας επιτόπου. Η Υπηρεσία Εξωτερικών Δράσεων είναι έτοιμη να αναλάβει συντονιστικό ρόλο σε συνεργασία με τι άλλε υπηρεσίε τη Ευρωπαϊκή Επιτροπή, να συμμετάσχουμε στι θεματικέ συζητήσει που θα διεξαχθούν στη Γενέβη που θα αναφερθούν στα κύρια θέματα του CRRF και να υπάρξει έτσι ένα πιο προβλέψιμο πλαίσιο για τη διεθνή συνεργασία και για θέματα που έχουν σχέση με την προστασία. Σε ό,τι αφορά τις πιλωτικές χώρες, στα πλαίσια του CRF, η Ευρωπαϊκή Ένωση είναι από τους πρώτους δωρητέ που συμβάλλει με συγκεκριμένε δράσεις, όπως για παράδειγμα στο πολιτικό πρόγραμμα με την Ουγκάντα. Για να γίνει η διαδικασία CRRF επιτυχία, χρειαζόμαστε την εμπλοκή και άλλων δωρητών και χωρών υποδοχής, σύμφωνα και με την διακήρυξη των Ηνωμένων Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Ευχαριστώ πολύ. Θα ακούσουμε τώρα τους ευρωβουλευτές που επιθυμούν να λάβουν το λόγο. Πρώτη κυρία Σράιν που συμμετείχε και στην αντιπροσωπεία που μετέβη στη Νέα Υόρκη. Έχεις ε, το λόγο. Ευχαριστώ. Κύριε Πρόεδρε, απευθύνω θερμό καλώς ορίσατε στους προσκεκλημένους μας σήμερα, γιατί για μας είναι, έχει κρίσιμη σημασία να παρακολουθήσουμε τη συζήτηση γύρω από το Global Compact, που βρίσκω ότι είναι πολύ σημαντικό να παραμείνει το Κοινοβούλιο, να εμπλακεί δηλαδή στη διαδικασία και να την παρακολουθεί. Έχω ένα πρώτο σχόλιο. Εκτιμώ την αισιοδοξία σας, αλλά είναι δύσκολο να θεωρήσουμε την Ευρωπαϊκή Ένωση ως πρωταθλητή της μετεγκατάστασης, γιατί ως γνωρίζετε οι χώρες μέλη δεν κατέσαν καν ικανές να υλοποιήσουν τις δεσμεύσεις που ανέλαβαν το 2015 σε ό,τι αφορά 160.000 με αντικαταστάσεις εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Και βέβαια πρώτα ε, την επανεγκατάσταση και μετά την μετεγκατάσταση και ούτω καθεξής. Ίσως ε, τα τελευταία νούμερα να τα γνωρίζουν της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, αλλά 20.000 περίπου relocations μιλούμε. Γι' αυτό, για τέτοιο, είναι λιγότερο από τα μισά από αυτά που είχαν υποσχεθεί. Και ταυτόχρονα ο Καναδάς, ένα παράδειγμα μόνο, κατέστησε 40.000 ανθρώπους τους τελευταίους μήνες. Άρα το πρόβλημα, το ευρωπαϊκό πρόβλημα δεν είναι ζήτημα αριθμών ή μέσων, αλλά είναι έλλειψη βούλησης. Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο κατ' επανάληψη έχει ζητήσει κατανομή των ευθυνών και να δημιουργηθούν νόμιμες οδοί πρόσβαση στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Αλλά το Συμβούλιο και δυστυχώς και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή τελευταία φαίνονται να μην ακούν και πολύ αυτά που λέμε εμείς στα ψηφίσματά μας. Ολοκληρώνω. Έχω μία ερώτηση. Πώς νομίζετε ότι η αλλαγή στο πολιτικό πλαίσιο και η νέα Αμερικανική διοίκηση θα ανατρέψει τις συζητήσεις για το Global Compact. Την ημέρα μετά από τη διάσκεψη κορυφής, ήμασταν και εμείς παρούσες εκεί, και η Αμερικανική κυβέρνηση είπε ότι θα αναλάβει συγκεκριμένε δεσμεύσεις. Αυτή η συζήτηση πώς προχωρεί τώρα μετά από την αλλαγή στην Αμερικανική κυβέρνηση και νομίζετε ότι θα επηρεάσει το συνολικό πλαίσιο των συζητήσεων σε ό,τι αφορά την ανάληψη συγκεκριμένων δεσμεύσεων. Και ένα τελευταίο σχόλιο. Αυτά που βλέπουμε είναι μια τάση δυστυχώς. Η ερώτηση μάλλον είναι πώς μπορεί να είναι συνεκτική η Ευρωπαϊκή Ένωση με τις δεσμεύσεις που ανέλαβε πέρυσι στη Νέα Υόρκη όταν όλες οι πολιτικές και οι προσπάθειες Συμβουλίου και Ευρωπαϊκής Επιτροπής φαίνεται να είναι προς την, προς, ε, μια προσπάθεια να μετατεθούν προς τα έξω τα σύνορα. Συμφωνία με την Τουρκία, συμφωνία με τη Λιβύη, συμφωνίες με αφρικανικές χώρες. Αν είναι σωστό αυτό που λέει η κυρία Χάνσεν, ότι 86% όλων των μετατοπισμένων και οι πρόσφυγες έρχονται από τον Νότο, νομίζω ότι με τον τρόπο αυτό διαπιστώνουμε ότι κινούμεθα στην αντίθετη κατεύθυνση. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ, Έλλη. Γεράρ Ντεπρέ. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Θα μιλήσω γαλλικά. Λέει ο κύριος Ντεπρέ. Άκουσα τις παρεμβάσεις σας με μεγάλο ενδιαφέρον. Το πρώτο λοιπόν που θέλω να ρωτήσω είναι το εξή. Έχετε μία δήλωση με μία ολοκληρωμένη απάντηση στο προσφυγικό ή τέλο πάντων προσπαθούμε να έχουμε αυτήν την ολοκληρωμένη απάντηση. Οπότε ρωτάω παγκοσμίω σε σχέση με αυτή την ολοκληρωμένη απάντηση και βλέποντας τα πράγματα έτσι όπως τα βλέπετε. Τι είναι αυτό που λείπει στην Ευρώπη για να έχει μια πραγματική πολιτική έτσι όπως καθορίζεται από την διακήρυξη της Νέας Υόρκης. Υπάρχουν κάποιοι τομείς στους οποίους πιστεύετε ότι έχουμε αδυναμίες, ότι κάτι θα έπρεπε να κάνουμε που δεν έχουμε κάνει. Δηλαδή από τη δικιά σας οπτική γωνία, ποιοι είναι οι τομείς εκείνοι στους οποίους θα πρέπει να βελτιώσουμε το έργο μας. Ξέρω ότι για την επανεγκατάσταση θα έπρεπε να βελτιώσουμε πολύ τις επιδόσεις μας, αλλά υπάρχουν και άλλα Έχουμε και άλλες αδυναμίες και άλλες σημεία στα οποία θα περιμένατε περισσότερο από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Και κάτι ακόμα πιο πρακτικό. Μιλήσατε για κάποιες χώρες που θα διευκολύνουν πιο πολύ την κατάσταση, θα είναι στην πρώτη γραμμή. Τι θα κάνουν δηλαδή, τι θα κάνουν αυτές οι χώρες, τι θα κάνει ο ΙΕ και τι περιμένετε από εμά. Προσπαθώ να καταλάβω στην πράξη έτσι, ποιος ακριβώς είναι ο μηχανισμός που βρίσκεται πίσω από την διαδικασία που περιγράψατε. Τέλος, είπατε ότι στο πρόγραμμα δράσης χρειάζονται περισσότερα μέσα. Η κυρία Χάντσεν το είπε. Περιμένετε περισσότερα μέσα από εμά. Πιστεύετε ότι η συνεισφορά των ευρωπαϊκών χωρών και όσον αφορά το Ευρωπαϊκό Ταμείο Ανάπτυξης και όσον αφορά τις πολιτικές που χρηματοδοτούμε στις διάφορες χώρες και την συμμετοχή μας όσον αφορά την υποδοχή προσφύγων, πιστεύετε ότι και εδώ βρισκόμαστε πίσω, ότι θα έπρεπε να κάνουμε περισσότερα για να σκούμε στο ύψος των ευθυνών μας. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ πολύ. Η κυρία Γκόμε. Καλώς ήρθατε και από μένα. Θα ήθελα πρώτα να δηλώσω ότι συμφωνώ απολύτως με την προλαλή Έλλη Σλάιν σε ό,τι αφορά τις δικές μας αντιφάσεις εδώ στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Και η ερώτησή μου προς εσάς έχει ως εξής. Πώς συμφιλιώνεται όλους αυτούς τους φιλόδοξους στόχους που έχουμε ανακοινώσει για το Global Compact και τα πράγματα που κάνουμε στην πράξη. Μόλις χθε, άλλοι χίλιοι άνθρωποι διεσώθησαν στη Μεσόγειο. Από 45.000 άτομα τα οποία έφτασαν μόνο φέτος στις ακτές Ευρωπαϊκής Υπήρου, θέτοντας βέβαια σε κίνδυνο τις ζωές τους, διότι δεν υπάρχουν ελεγχόμενες νόμιμες οδοί, εκτός βέβαια από τις ε, οδές, τι ελεγχόμενες από τους διακινητές για να έρθουν στην Ευρώπη. Διότι η Ευρώπη ε, δεν ανοίγει νόμιμες ασφαλείς οδούς. Δεν νομίζετε ότι θα είναι αυτό ένα κρίσιμο ερώτημα που θα πρέπει να συμπεριλάβετε στα σχόλιά σας προς την Ευρωπαϊκή Ένωση όπως η νόμιμη οδός που έχει ανοίξει ο Καναδάς. Και επίσης το μήνυμά σας προς τους Ευρωπαίους αντιλαμβάνομαι ότι χρειάζεστε ε, κονδύλια, πολιτική στήριξη, αλλά η ίδια η διαδικασία δεν διασώζεται εάν δεν επιφέρει κάποια σημαντική διαφορά για τους ανθρώπους που επιδιώκεται να στηρίξετε, ιδίω τους πρόσφυγες. Μπορεί λοιπόν η Ευρώπη πράγματι να τηρήσετε επισημένα σε ό,τι αφορά την προστασία των προσφύγων εάν επαναλάβει την ίδια παράνομη και ανήθικη συμφωνία που έχει με την Τουρκία τώρα με την Λιβύη όπου εσείς ως αρμοστής δεν έχετε προσωπικό δεν έχετε καν νομικό καθεστώς στη Λιβύη και προφανώς η πρόθεση της Ευρωπαϊκής Ένωσης είναι να αναθέσει εξωτερικά ας πούμε αυτό το πράγμα το οποίο αποκαλεί προστασία μεταναστών και προσφύγων. Να τα αναθέσει εξωτερικά, δηλαδή σε εσά. Μπορείτε ναι, όμω εσεί να αναλάβετε το έργο αυτό σε μια χώρα όπω η Λιβύη. Τέλος, μπορούμε να αντιμετωπίσουμε την προστασία των προσφύγων με σοβαρό τρόπο εάν συνεχίσουμε να αγνοούμε το κρίσιμο πολιτικό θέμα που βρίσκεται στο επίκεντρο δεν είναι καθαρά ανθρωπιστικό, είναι και πολιτικό το θέμα, όπως άλλωστε το δέχτηκε και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Και χρειάζεται τέτοια προσέγγιση. Και βεβαίως να έχει και αναπτυξιακή διάσταση. Εγώ συγκλονίστηκα πραγματικά από την ομιλία του Γενικού Γραμματέως των ΗΠΑ του κ. Κουτέρες, που εξεφώνησε στην Άντι Σάβεμπα τον Ιανουάριο, όταν επισκέφθηκε την πόλη για το θέμα των προσφύγων. Γνωρίζω ότι η χώρα μας έχει, ότι η χώρα αυτή μάλλον έχει υποστηρίξει πολλούς πρόσφυγες από άλλες γειτονικές της χώρες, αλλά παράγει και πολλούς πρόσφυγες λόγω των καταπιστικών πολιτικών της. Μήπως όλοι κοροϊδεύουμε τους εαυτούς μας αν συνεχίσουμε να παραγνωρίζουμε αυτό το κρίσιμο θέμα κυβερνήσεων οι οποίες δρούν με καταπιστικό τρόπο και προκαλούν έτσι πρόσφυγε ή προσφυγικά ρεύματα. Αν πάτε στο Καλέ θα βρείτε εκεί πολλούς πρόσφυγες από την Αιθιοπία. Ευχαριστώ. Άννα. Σας ευχαριστώ, Κλόντ. Και εγώ χαίρομαι για το γεγονός ότι έχουμε αυτή την ευκαιρία να ακούσουμε πώς προχωρούν τα πράγματα και οι εργασίες ε, όσον αφορά αυτή τη νέα δήλωση, διακήρυξη της Νέας Υόρκης. Θα ήθελα να θυμίσω και στους, και στους φιλοξενούμενους μας ότι πριν από ένα χρόνο ακριβώς εδώ σε αυτό το κοινοβούλιο ε, με μεγάλη πλειοψηφία υπερψηφίσαμε ένα ψήφισμα που αφορά σχεδόν όλα όσα θέλουμε να ε, όσα μάλλον συμπεριλαμβάνονται και στη διακήρυξη της Νέας Υόρκης. Και ο τόνος ήταν η αρχή της αλληλεγγύης, δηλαδή μεταρρύθμιση του Δουβλίνου, σύστημα μόνιμης ανακατανομής, που το οποίο θα είναι μονίμως δεσμευτικό, ε, η ενεργοποίηση των ε, ανθρωπιστικών αποστολών, πολιτική ένταξη και ενέργειες για τα, τα αίτια της μετανάστευσης. Εάν κανείς κλείσει τα μάτια θα έλεγε ότι όλα πάνε χαρά. Πάνε μια χαρά ότι είμαστε τέλεια, γιατί έχουμε γράψει πράγματα που πραγματικά θέλουμε να γίνουν. Όμω τώρα πρέπει να δούμε αν, αν έχουν υλοποιηθεί όλα αυτά ή όχι. Αλλά προ μεγάλη μου έκπληξη, εγώ βλέπω ότι μετά από ένα χρόνο από αυτή τη διακήρυξη, όχι και με τόση έκπληξη, ότι συνεχίζουμε να συζητάμε αν θα πρέπει όλα αυτά να εφαρμοστούν ή όχι. Και κυρίω βρισκόμαστε ενώπιον τη πραγματικότητα που ήδη είχαμε διαπιστώσει επί τόπου. Όπω, α πούμε, οι πανεγκαταστάσει, οι μετεγκαταστάσει, η οικογενειακή επανένωση, η δουλειά, η κατάσταση στι χώρε επιστροφή. Τα ξαναβρίσκουμε πάλι τα ίδια θέματα. Μα πότε θα τελειώσει αυτή η κατάσταση. Τα γνωρίζουμε ότι πρέπει να τα κάνουμε όλα αυτά. Δεν είναι καινούρια. Ναι, υπάρχει πολιτική κρίση πολύ έντονη, κρίση ελληνικής, γιατί πολλές από τις προτάσεις τις γνωρίζουμε. Αλλά επικρατεί και μεγάλη υποκρισία, γιατί αν δούμε ας πούμε την περίπτωση της Λιβύης, όπου αν αρχίσουμε να μιλάμε για ε, για επανεγκατάσταση στη Λιβύη και να επιστρέφουμε κόσμο στη Λιβύη, μα πώς μπορούμε να συμφωνήσουμε να συμφωνήσουμε να επιστρέφονται άνθρωποι εκεί σε αυτά τα στρατόπεδα συγκέντρωσης που τα γνωρίζουμε όλοι. Για το Τζιμπουτί επίσης γνωρίζουμε τι συμβαίνει. Ε, υπάρχουν πρόσφυγες από την Ιεμένη. οι οποίοι δεν μπορούν καν να μπορούν να εγκατασταθούν σε άλλη χώρα. Γιατί το Τζιμπουτί χρησιμοποιείται ως μοντέλο για να μπορέσουν να εγκατασταθούν και να ενσωματωθούν εκεί. Δεν ε, τους προσφέρεται καν η δυνατότητα να πάνε αλλού. Αντίθετα, τους δίνεται ένα έγγραφο παραμονής που τους εμποδίζει ούτε καν να πούν ε, τι θέλουν και ότι θέλουν να πάνε αλλού και να εγκατασταθούν αλλού. Εγώ ρωτώ αν το γνωρίζετε αυτή την κατάσταση. Το τελευταίο θέμα είναι το πολιτικό θέμα που έθιξε η Άννα. Όταν μιλάμε για ε, μετεγκαταστάσεις, και έχουν γίνει τις περισσότερες φορές εκτός των δικών μας συνόρων. Μιλάμε και για χώρες οι οποίες υποτίθεται είναι ασφαλείς, χωρίς να λαμβάνουμε υπόψη όμως την παραβίαση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, ούτε την πολιτική κατάσταση. Και διερωτώ κατά πόσο όλα αυτά λαμβάνονται υπόψη στο πλαίσιο αυτής της διακήρυξης της Νέας Υόρκης. Ευχαριστώ. Thank you, Ευχαριστώ, Σεσίλ. Γιώργο. Ευχαριστώ πολύ και ευχαριστώ τους προσκεκλημένους μας που ήρθαν. Όπως γνωρίζετε, το είπαν και οι συνάδελφοι, εργαζόμαστε σε διάφορα επίπεδα προκειμένου να πετύχουμε μια όσο γίνεται πιο ολοκληρωμένη προσέγγιση. Εγώ είμαι η συγγήτρια έκθεσης όσον αφορά το πρόγραμμα επανεγκατάστασης και προσπαθούμε εδώ με τους συναδέρφους στην Επιτροπή μας ε, να καταστήσουμε το κείμενο όσο γίνεται καλύτερο. Είναι σαν να μην έχει αποφασίσει η Ευρωπαϊκή Ένωση τι δρόμο θα ακολουθήσει, κατά πόσο θα σταματήσει να εξωτερικεύει τα σύνορά της και να αποσύρεται από τις δεσμεύσεις που έχει πάρει μέχρι τώρα ή όχι. Είναι σαφές όμως ότι περισσότεροι εδώ ξανά και ξανά έχουμε πει ότι θέλουμε να κάνουμε αυτό που κι εσείς θέλετε, δηλαδή να αναλάβουμε τις ευθύνες μας. Τώρα, επειδή είμαι συγκήτρια για την επανεγκατάσταση, θέλω να πω ότι η επανεγκατάσταση είναι μόνο ένα κομμάτι του παζλ. Υπάρχει η επανένωση οικογενειών και άλλα. Η ασφαλής ε, οδή για τη μετανάστευση κλπ. Η δικιά μας η φιλοδοξία στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και συνεργαζόμενοι εδώ και με τους συναδέρφους είναι να έχουμε ένα πιο φιλόδοξο πρόγραμμα από αυτό το οποίο ήδη προτείνεται. Θέλω από αυτού το δικό σας ε, το σχόλιο. Θέλουμε να αυξήσουμε τα νούμερα, θέλουμε να αυξήσουμε την ποιότητα και θέλουμε να αλλάξουμε και το μήνυμα. Γιατί ναι, η Ευρωπαϊκή Ένωση μπορεί να παίξει σημαντικό ρόλο. Και αν δεν το κάνουμε αυτό με την επαναγκατάσταση, θα αποτύχουμε και στο μήνυμα που στέλνουμε. Υπάρχει το σχέδιο πάντως της εκθεσής μου και θα ήθελα τα δικά σας σχόλια από αυτού. Η ύπατη αρμοστία του ΟΗΕ για τους πρόσφυγες έχει πολύ σημαντικό ρόλο να παίξει. Συγχρόνως όμως και η Ευρωπαϊκή Ένωση συνολικά θα έπρεπε να σταθεί στο ύψο τη και να συνεργαστεί μαζί σας για να έχουμε καλύτερα αποτελέσματα. Θέλω να ακούσω για εσά τι γεωγραφικές προτεραιότητες υπάρχουν. Γιατί όπως είπαν και οι συνάδελφοι θα ήταν λάθος αν αρχίζαμε τώρα να έχουμε τέτοια προγραμματάκια με τρίτες χώρες. Πρέπει να είμαστε σίγουροι ότι γίνεται η ανθρωπιστική βοήθεια, ότι υπάρχει. Και θα ήθελα να συνδέσουμε τα ευρωπαϊκά προγράμματα με το συνολικό πρόγραμμα επανεγκατάστασης. Θέλω λοιπόν και από αυτού τα σχόλιά σας και παρακαλώ ότι άλλες ιδέες έχετε και στο μέλλον να επανέλθετε. Ευχαριστούμε. Τέλος Μπάρμπαρα Σπινέλη. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Έχω κάποιες ερωτήσεις και ευχαριστώ τον, τους εκπροσώπους ε, της ΥΠΑ του ΟΗΕ επειδή είστε σήμερα εδώ αλλά θέλω να ρωτήσω κάποια πράγματα για το λεξιλόγιο που χρησιμοποιείτε σε αυτό το παγκόσμιο σύμφωνο γιατί οι λέξεις είναι σημαντικές και ορισμένες από αυτές που χρησιμοποιήθηκαν είτε δεν είναι απόλυτα σαφείς είτε κάποιες φορές παραμένουν απλά εφημισμοί κατά τη γνώμη μου. Κάτι λοιπόν που θα ήθελα πολύ να γνωρίζω είναι ακριβώς τι σημαίνει όταν λέτε self-reliance, δηλαδή ε, η αντοχή του ίδιου του πρόσφυγα ε, η εμπιστοσύνη στον εαυτό του. Τι ακριβώς εννοείται, γιατί υπάρχει συνέχεια στο κείμενο. Κάτι ακόμα λέγεται εδώ ότι θα βοηθηθούν οι χώρες που ε, φιλοξενούν τους πρόσφυγες. Θα στηριχτούν δηλαδή ή θα βελτιωθούν οι συνθήκες στις τρίτες χώρες. Και εδώ υπάρχει και ο εφημισμός που λέει ότι θα μοιραστούν πιο ισότιμα οι ευθύνε. Εγώ πιστεύω ότι ένα πιο σαφές, μια πιο σαφή γλώσσα θα έπρεπε να περιλαμβάνει και μια πιο έντονη δέσμευση κατά της έλλειψης ισορροπίας, της βαθιάς, βαθύτατης παγκόσμια έλλειψη ισορροπίας που υπάρχει ανάμεσα στο βορρά και στο νότο και τα στοιχεία που δίνεται είναι 86% των προσφύγων βρίσκονται στο νότο του κόσμου. Μα τότε πρέπει να μιλήσουμε για μια έλλειψη ασυσορροπίας που θα πρέπει να διορθωθεί και όχι απλά για στήριξη των χωρών που δέχονται τους πρόσφυγες. Κάτι ακόμα αφορά τους επαναπατρισμούς. Και εδώ δεν έχω καταλάβει πολύ καλά τη γλώσσα πάλι. Λέγεται για επαναπατρισμό, returns, βιώσιμους και θελοντικούς επαναπατρισμούς. Μα γνωρίζετε καλά ότι συμφωνίες με κάποιες τρίτες χώρες, ιδιαίτερα το Αφγανιστάν, προβλέπουν αναγκαστικούς επαναπατρισμούς. Οπότε δεν καταλαβαίνω και πολύ καλά. Ακόμα και για ε, ανήλικους, μη ασυνόδευτους ανήλικους ε, καταναγκαστικοί επαναπατρισμοί. Εσείς πώς μιλάτε λοιπόν ε, για την Ευρώπη, λες και είναι ο πρωταθλητής στον κόσμο και έπειτα αυτή την πολιτική του μηνύματος που λέτε, το messaging. Χαίρομαι για το γεγονός ότι αναγνωρίζετε ότι υπάρχει ανάμεσα στους πρόσφυγες και τους οικονομικούς μετανάστες πρόβλημα. για να διαχωρίσουμε, να κάνουμε διάκριση μεταξύ τους, αλλά ξέρετε ότι στις διάφορες ευρωπαϊκές χώρες γίνεται αυτός ο διαχωρισμός παρόλα αυτά και ότι εν γέννη γίνεται λόγος για περισσότερους οικονομικούς μετανάστες και άρα για πολιτικές επαναπατρισμού που θα πρέπει να γίνουν, να υλοποιηθούν μαζικά. Και έπειτα, ετήσιες διαβουλεύσεις που λέτε ότι θα κάνετε με τις ΜΚΟ. Και εδώ, σε αυτή την περίπτωση, γνωρίζετε ότι η ΜΚΟ είναι υπό πολύ σοβαρή επίθεση. Πολλές ΜΚΟ που κάνουν ειδικά έρευνα και διάσωση κυρίως στο ιδιόργα της Σικελίας αλλά και κοντά στη Λιβύη και ότι η κοινή γνώμη πολύ φοβάται από την από τα όσα λέγονται για τις ΜΚΟ στην Ευρώπη, ότι δηλαδή λειτουργούν ως pull factor ε, για τη Λιβύη. Και εδώ δεν μου φαίνεται να είναι και πολύ πρωταθλήτρια η Ευρώπη. Σας ευχαριστούμε πολύ. Λοιπόν, ακούσατε τις ερωτήσεις και έχω και μία τελευταία εγώ. Είχαμε μια συνάντηση πολύ ενδιαφέρουσα, σίγουρα, αλλά οσον αφορά το Παγκόσμιο Σύμφωνο, η κυρία Μπιόργκο το έθεσε πολύ σωστά. Ένα από τα προβλήματα που έχουμε είναι ακριβώς η έλλειψη εφαρμογής, γιατί έχουμε πολιτικές, για την επανακατάσταση, τη μετεγκατάσταση. Τα έχουμε όλα αυτά. Δεν είναι θέμα πολιτικής, είναι θέμα εφαρμογής και έλλειψης πολιτικής βούλησης πολλές φορές, όπως είπε και η κυρία Κέγκε. Συνεπώς, η ερώτησή μου είναι για το Παγκόσμιο Σύμφωνο. Θα έχουμε τον Γενικό Γραμματέα του ΕΕ την επόμενη εβδομάδα σε μας. Δεν πρόκειται για ένα δεσμευτικό μέσο, έτσι. Οπότε απαιτεί στήριξη. Αλλά πριν από αυτό απαιτείται γνώση. Ο κόσμος λοιπόν το γνωρίζει είναι ενήμερος για αυτή την προσπάθεια και πώς εμείς μπορούμε να παίξουμε ρόλο έτσι ώστε τα προβλήματα τα δικά μας που είναι η αντίσταση, η μη εφαρμογή να μην υπάρξουν και εδώ όσον αφορά το παγκόσμιο αυτό σύμφωνο κυρίως όσον αφορά την επανεγκατάσταση που είναι σίγουρα μια αποτυχία. Ευχαριστώ. Η κυρία Χάνσεν, νομίζω ότι υπάρχουν πολλά σχόλια. Ε, θα μπορούσα σε όλα να σχολιάσω, αλλά δεν γίνεται. Θα απαντήσω εγώ σε μερικά και ο κύριος Μπάλτη σε κάποια άλλα. Λοιπόν, ποια είναι η καρδιά του ζητήματος, ο πυρήνας του ζητήματος. Κατά πόσο οι χώρες μέλη πρέπει να κάνουν κάτι παραπάνω και αν η Ευρωπαϊκή Ένωση μπορεί να κάνει κάτι παραπάνω. Και αυτό το είπα όταν αναφέρθηκα στην επανακατάσταση. Γιατί είναι αλήθεια ότι σε αυτό το τομέα δεν θα λέγαμε ότι είναι η Ευρώπη. Όχι. Πιστεύουμε ότι μπορούν να γίνουν πολύ περισσότερα για την επανεκατάσταση. Πιστεύουμε ότι μπορούν να γίνουν περισσότερα και όσον αφορά την επανένωση οικογενειών. Πιστεύουμε ότι είναι πολύ σημαντικό για τα κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης να διαφοροποιήσουν τις ποσοστώσεις τους όσον αφορά την επανεγκατάσταση, ώστε να ανταποκρίνεται και το πλαίσιο για την επανένωση οικογενειών στις πραγματικές ανάγκες. Δηλαδή να βασιστούμε εδώ πέρα περισσότερο στις πραγματικές ανάγκες των προσφύγων, καταρχήν. Πιστεύουμε ότι επιπλέον από την επανεγκατάσταση είναι αναγκαία η επανένωση. Είπα ότι εδώ μπορούν να γίνουν πολύ περισσότερα. Και τώρα το θέμα της διευκόλυνσης της επανένωσης αυτής είναι ένας τομέας όπου επίσης μπορούν να γίνουν περισσότερα και θα πρέπει να προσεχθεί όλος ιδιαίτερος. Να εντοπιστούν και οι ευκαιρίες που υπάρχουν προκειμένου να διευκολύνεται η επανένωση των οικογενειών. Θα έκανε έκκληση μάλιστα και στα ευρωπαϊκά θεσμικά όργανα σίγουρα να στηρίξουν επιπλέον διόδους αποδοχής προσφύγων και μεταναστών. Τώρα λίγο να έρθω στο πολιτικό πλαίσιο. Με ρωτήσατε κατά πόσο έχει αλλάξει και κάποιος αναφέρθηκε και στην τελευταία διάσκεψη με τον Γενικό Γραμματέα, τον Πρόεδρο Ομπάμα και κάποιες χώρες που φιλοξενούν πρόσφυγες. Υπήρξαν δεσμεύσεις και από πλευράς Ευρωπαϊκής Ένωσης αλλά και από πλευράς των ε, χωρών. Πολλοί ρωτούν τι θα μπορούσαμε να κάνουμε να είμαστε θετικοί πρώτα απ' όλα. 500.000 παιδιά πάνε σχολείο στην Τουρκία και αυτό με τη βοήθεια πόρων από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Και υπάρχουν πολύ περισσότεροι πρόσφυγες που έχουν πρόσβαση σε ένα νοικοκυριό, σε δουλειά. Υπάρχουν λοιπόν και τα θετικά. Σίγουρα το πολιτικό πλαίσιο είναι δύσκολο. Δεν είμαστε πολιτική οργάνωση, αλλά παρατηρούμε και εμείς τι γίνεται με τις εκλογές ανά τον κόσμο, με ιδιαίτερο ενδιαφέρον. Και υπάρχουν εξελίξεις που είναι ανησυχητικέ. Όσον αφορά τη γλώσσα που χρησιμοποιεί κανείς για την μετακίνηση αυτή των προσφύγων και για την αντιμετώπιση τους, πώς θα τους προστατεύσουμε. Εμείς δεν πιστεύουμε ότι η προστασία των προσφύγων είναι σε αντίθεση με την ασφάλεια των διαφόρων χωρών. Δεν πιστεύουμε ότι υπάρχει μια τέτοια αντίφαση εδώ. Είναι συμβατά και τα δύο. Όσον αφορά το Γενικό Γραμματέα και την επικείμενη επίσκεψή του στο Στρασβούρο, φυσικά δεν μπορώ να προκαταλάβω τι θα πει, αλλά επειδή ήταν ε, πρωθυπουργός στην ε, Πορτογαλία και ήταν, έχει περάσει και από την ε, πατερμοστή για τους πρόσφυγες, γνωρίζει τα πράγματα καλά και τίποτα παραπάνω δεν τον απασχολεί στη θέση που είναι από την ε, προληπτική διπλωματία. Σίγουρα η συνεισφορά του θα είναι ιδιαίτερα πολύτιμη. Το θέμα των ποσοστών είναι κάτι πολύ σημαντικό ξέρουμε από την έγκαιρη προειδοποίηση ότι με την κατάλληλη ρύθμιση και νομοθεσία μπορούν να αποφευθούν μετακινήσεις πληθυσμού όσον αφορά τώρα την εφαρμογή των πολιτικών. Ένας από τους λόγους για τους οποίους πιστεύουμε ότι είναι σημαντική η διακήρυξη της Νέας Υόρκης είναι επειδή επαναλαμβάνει την δέσμευση υπέρ της σύμβασης για τους πρόσφυγες Βέβαια, όπως και οπουδήποτε αλλού συμβαίνει και εδώ η διακήρυξη αυτή θα αποδειχτεί καλή εφόσον μπορεί να εφαρμοστεί στην πράξη. Να υπάρχει δηλαδή ένα νομικό πλαίσιο που να λειτουργεί. Και το ίδιο μπορούμε να πούμε και για την μετανάστευση. Εκεί βέβαια δεν έχουμε προχωρήσει τόσο πολύ, αλλά υπάρχουν και εδώ ανθρώπινα δικαιώματα, τα οποία πρέπει να υπενθυμίζουμε ότι ισχύουν παγκοσμίω και για τους μετανάστες. Χρηματοδότηση τώρα. Η χρηματοδότηση αποτελεί μια ανησυχία για μα. Και όταν μιλάμε για μια χώρα σαν την Ουγγάντα, για παράδειγμα, η οποία τα κάνει όλα καλά όσον αφορά την προοδευτική τη πολιτική για του πρόσφυγε, ανοίγει την αγορά εργασία, τη του δίνει γη, εκπαίδευση, έχει σχεδιασμό στην ομοθεσία κτλ. Δεν χρηματοδοτείται όμω επαρκώ. Και όχι, δεν στρεφόμαστε στην Ευρωπαϊκή Ένωση για να ζητήσουμε λεφτά, ούτε στι χώρε μέλη για την Ουγγάντα. Σίγουρα είσαστε όλοι πολύ σημαντικοί δωρητές. Μια κρίση αλληλεγγύης τώρα. Είναι ένας όρος που χρησιμοποίησε ο προηγούμενος Γενικός Γραμματέας. Δεν ε, πιστεύουμε ότι υπάρχει κρίση αριθμών, υπάρχει κρίση αλληλεγγύης. Με αυτό συμφωνούμε. Οπότε είναι θέμα διαχείρισης της κατάστασης και όταν μιλάμε για ένα εκατομμύριο ανθρώπους που ήρθαν το 2015, όπου στην Ευρώπη έχουμε ένα πληθυσμό 500 εκατομμύρια και το συγκρίνουμε αυτό με το Λίβανο, όπου ένα στους πέντε είναι πρόσφυγας, ε, προφανώς πιστεύουμε ότι αν υπάρχει πολιτική βούληση υπάρχει και ο τρόπος. Δεν θέλω τώρα να μπω στη συζήτηση για τη Λιβύα. Δεν είμαι η κατάλληλη, αλλά υπάρχουν θέματα ασφάλειας. Και είμαστε ενήμεροι. Και υπάρχει θέμα δηλαδή με την επιστροφή ανθρώπων σε μια χώρα όπως η Λιβύη, όπου δεν υπάρχει επαρκής προστασία και χρειάζονται και ανθρωπιστική βοήθεια οι άνθρωποι που βρίσκονται εκεί. Οπότε η κατάσταση νομίζω ότι μιλάει από μόνη της όσον αφορά τη Λιβύη. Τώρα για το θέμα των ορισμών και για τις πιλωτικές χώρες που θα συμμετάσχουν, μάλλον για τις χώρες που θα συμμετάσχουν πιλωτικά. Ίσως να δώσω το λόγο στον κύριο Μπάλτη. Σας ευχαριστώ πολύ πάντως για τον προβληματισμό σα. Είστε ειλικρινεί και αυτό είναι πάντα, αυτό ισχύει πάντα και χαίρομαι γι' αυτό. Και παρά λοιπόν το δικό σας τον προβληματισμό, απόλυτα θεμητός, θα συνεχίσουμε να έχουμε τα μάτια στραμμένα στην Ευρώπη για πολιτική και παγκόσμια ηγεσία. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ πολύ. Για να μπορέσω να κάνω κάποιες συμπληρωματικές παρατηρήσεις από τις διάφορες ευθείες ερωτήσεις και παρατηρήσεις που κάνατε, σημειώνουμε ίσως δύο μηνύματα. Πρώτο, κάνουμε αρκετά. Απάντηση όχι, δεν κάνουμε αρκετά όλοι μας. Θα έπρεπε να κάνουμε περισσότερα πράγματα, διότι υπάρχουν μεγάλες ανάγκες και δεν είναι μονάχα η προσπάθεια να εξεύρουμε λύσεις στα προβλήματα των προσφύγων, αλλά να δούμε και ποια είναι τα αίτια στη βάση τους, οι ρίζες. Υπάρχουν θεσμοί, υπάρχουν φορείς που είναι σε καλύτερη θέση να εξετάσουν τις ρίζες των προβλημάτων, καθώς και τις συνθήκες που μπορούν να φέρουν στους ανθρώπους να έχουν λιγότερη ανάγκη διεθνούς προστασίας. Λοιπόν, δεν κάνουμε απαραίτητα αρκετά. Κάνουμε ορισμένα πράγματα. Πιστεύω ότι οι άνθρωποι ανταποκρίνονται και οι εκπρόσωποι των κυβερνήσεών σας σε σχέση με ορισμένες χώρες. Βλέπουμε πρόσβαση στην εκπαίδευση, βλέπουμε καταχώρηση βελτιωμένη, αυξανόμενη. Βλέπουμε στήριξη εταίρων και οικονομική βελτιωμένο επίπεδο προστασίας σε πολλές χώρες και μετακίνηση πολιτικών από τις θέσεις που είχαν παλαιότερα. Και δεν είναι μονάχα χρηματοδότηση, είναι και πολιτική στήριξη. Ναι, λοιπόν, νομίζω ότι πρέπει πράγματι να κάνουμε περισσότερα από όσα κάνουμε. Εσείς παίζετε ένα σημαντικό ρόλο στην ανταπόκριση της ε, ανάγκης αυτές. Έγιναν και ερωτήσεις σχετικά με το τι χρειαζόμαστε στο ευρωπαϊκό επίπεδο. Νομίζω ότι είναι θεμητή ερώτηση. Και νομίζω ότι εμείς εδώ αναφερθήκαμε σε δύο τομείς όπου μπορεί να βελτιώσει τη δράση της Ευρώπη. Αύξηση του αριθμού των θέσεων επανεγκατάστασης και οι χώρες που αποδίδουν μεγαλύτερη σημασία στην επανεγκατάσταση είναι οι Ηνωμένε Πολιτείε. Και γνωρίζετε ότι έγιναν σοβαρότατε αλλαγέ στο επίπεδο αυτό. Δεν ζητούμε από την Ευρώπη να κάνει πράγματα που δεν μπορεί ή πάντω δεν μπόρεσε για μεγάλο διάστημα. Ζητούμε πάντω να υπάρξει αύξηση των αριθμών. Και αυτό είναι το μήνυμα που περνούμε. Είτε πρόκειται για κεφάλαια, είτε πρόκειται είτε πρόκειται, συγγνώμη, είτε πρόκειται για τις πρωτεύουσε, είτε πρόκειται για τους θεσμούς. Να υπάρξει μεγαλύτερη στήριξη, μεγαλύτερη αριθμό ανθρώπων που να έχουν την ελπίδα ότι θα επανεκατασταθούν, ότι θα επανενωθούν με τις οικογένειές τους. Αυτό θα μας βοηθήσει όλους να τους εμποδίσουμε τους ανθρώπους αυτούς να λάβουν πάρα πολύ επικίνδυνες αποφάσεις όπου πραγματικά πολλοί άνθρωποι θα χάσουν τη ζωή τους και στη Μεσόγειο ή και στον Περσικό κόλπο ή και προς τον νότο της Αφρικής, γιατί έχουμε και αυτό το πρόβλημα, και την Ασία βεβαίως και αλλού. Μπορούμε να κάνουμε λοιπόν περισσότερα πράγματα, ναι. Εκεί μπορούμε να κάνουμε περισσότερα πράγματα. Εάν μπορώ να επανέλθω στα παραδείγματα που αναφέρατε, όπως ο Καναδάς, μπορούμε να προσβλέπουμε σε παραδείγματα όπως αυτές οι χώρες και ήθελα επίσης να με επιτρέψετε να κάνω μια διόρθωση. Δεν νομίζω ότι οι πρόσφυγες στην Ιεμένη παρεμποδίζονται από την επανεγκατάσταση. Είναι πολύ περιορισμένη οι διαθεσιμή χώρη Καμιά εθνότητα, καμιά εθνικότητα δεν παρεμποδίζεται από το να επανεγκατασταθεί. Εξετάζουμε όμως τους όρους, τις συνθήκες υπό τις οποίες χορηγεί το άσυλο. Και δεν είναι όλες κατάλληλες ή δεν έχουν όλες την ταχύτητα που θα θέλαμε. Μπορείτε να έχετε κάποια πρόσωπα τα οποία κατευθύνονται στην επανεγκατάσταση και να χρειάζονται δύο ή τρία χρόνια για ορισμένες χώρες. Πιστεύουμε λοιπόν ότι δεν υπάρχουν καταστάσεις που αποτρέπουμε κάποιες εθνικότητες από το να επαναγκατασταθούν, εκτός πλέον αν δεν υπάρχουν λόγοι που να επιτρέπουν πλέον το χαρακτηρισμό τους ως προσφύγων. Και αυτά που είπατε για τον Τζιμπουτή είναι αλήθεια. Και ήταν ενδιαφέρον που άκουσα για τις θετικές πολιτικές τις οποίες αναφερθήκατε. Νομίζω κυρία Σεσίλ έχουμε ετήσιες τριμερείς διαβουλεύσεις για την επανεγκατάσταση με χώρες προς τις οποίες κατευθύνεται η επανεγκατάσταση και με τις χώρες αυτές μπορούμε να κάνουμε και άλλες συζητήσεις για να υπάρξουν συμπληρωματικές δράσεις. Έγιναν και ερωτήσεις σχετικά με την δυνατότητα να βασίζονται τα άτομα στις δυνάμεις τους. Self-reliance. Ορισμένα άτομα δεν ζητούν βοήθεια. Αυτό που χρειάζονται είναι να τους δοθεί ένα περιβάλλον στο οποίο να μπορούν να ζήσουν σε αξιοπρέπεια. Με ανεξάρτητο τρόπο, όπως εσείς και εγώ και αυτό μπορεί να γίνει στη βάση μιας οικονομικής δραστηριότητας ή ελευθερίας κίνησης ή και τη δυνατότητα του επιχειρήν. Αυτή η αρχή της εξάρτησης από τις δικές σου δυνάμεις που επιτρέπουν στον πρόσφυγα να ζήσει με τις δικές του δυνάμεις ανεξάρτητος και βεβαίως εκεί να ληφθούν υπόψη ο εθελοντικός επαναπατρισμός, η επανεγκατάσταση ή η τοπική ενσωμάτωση. Αυτά είναι τα βασικά μηνύματα. Έγινε και μια ερώτηση σχετικά με την ίδια τη διακήρυξη της Νέας Υόρκης. Κύριε Πρόεδρε, νομίζω ότι εσείς είστε σε θέση να μας βοηθήσετε περισσότερο. Παρόλο που το κείμενο αυτό δεν έχει δεσμευτικό χαρακτήρα, η προστασία των προσφύγων και των ανθρώπων που βρίσκονται σε ανάγκη στήριξης είναι συχνά σημαντική προσπάθεια, επίπονη αλλά και οδυνηρή και νομίζω ότι με κάποια στήριξη από εσά μπορούμε να κάνουμε και την διακήρυξη αυτή της Νέας Υόρκης ένα συμπληρωματικό έγγραφο το οποίο θα βοηθήσει και στην εφαρμογή πιο δεσμευτικών διακήρυξεων όπως το 1951. Σας Ευχαριστώ, λέει ο Πρόεδρο, και εγώ σα ευχαριστώ που ήρθατε σήμερα εδώ. Έχουμε μόνιμε και διαρκεί σχέσει μαζί σα και όπω καταλάβατε και από τη συζήτηση, δεν υπάρχει έλλειψη επαφή με την πραγματικότητα. Έχουμε ε, ανθρώπου που είναι εμπειρογνώμονε, έχουμε ε, κατανόηση, γνωρίζουμε ακριβώ ποια είναι τα προβλήματα. Αυτό που θέλουμε να καταστήσουμε απόλυτα σαφέ είναι ότι συμφωνούμε μαζί σα ε, στην πορεία ήδη με του συντονιστέ έχουμε προτείνει σωστή και λεπτομερή ε, παρακολούθηση της διαδικασίας της διακήρυξης ε, της ε, Νέας Υόρκης μέχρι το Σεπτέμβριο του 2018 του 2016 έχουμε έρθει σε επαφή με τους ηθήνοντες της υπηρεσίας εξωτερικής δράσης, με τους συναδέλφους της DigiHome και συμμετέχουμε σε συνεδριάσεις κλειδιά, οπότε παρακολουθούμε στενά την διαδικασία, το διάλογο της, ε, του ΙΠΑ του αρμοστή για τους πρόσφυγες, ε, τις διεθνείς ε, σχετικές συνελεύσεις. Προσπαθούμε λοιπόν να έχουμε αυτή την συμμετοχή, συνεργαζόμαστε στενά με τους συναδέλφους της, εξωτερικής, της Υπηρεσίας Εξωτερικής Δράσης και με τις άλλες επιτροπές μας εξωτερικών υποθέσεων και ανάπτυξης. Ελπίζω λοιπόν ότι οι συνάδελφοι της ε, ΙΑΔ θα μας βοηθήσουν στα επόμενα βήματα. Σας ευχαριστώ και πάλι για την υψηλή ποιότητα της απόψινής συζήτησης. Ε, συνάδελφοι και συνάδελφοι από την ΥΠΑ τη Αρμοστία και ε, τώρα πρέπει να προχωρήσουμε στο επόμενο μας θέμα. Καθώ um, Καθώς αποχωρούν λοιπόν οι προσκεκλημένοι μας, ε, θα πάμε στο σημείο 4, γιατί έχουμε ελαφρώς καθυστερήσει, αλλά πιστεύω πως άξιζε, γιατί ε, πολλοί συνάδελφοι ήθελαν να λάβουν μέρος στη συζήτηση. Περνάμε λοιπόν στο σημείο 4 που είναι ο δρόμος ε, να προχωρήσουμε για τα θέματα τα μεταναστευτικά ε, Αφγανιστάν και Ένωση. Το σχετικό πρόγραμμα το αποκαλέσαμε κοινή πορεία εμπρός και εδώ στι 14 Νοεμβρίου οι συντονιστέ αποφάσισαν να ζητήσουν συμβουλέ από την νομική υπηρεσία σε σχέση με αυτήν την συμμετοχή του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου σε αυτή την κοινή πορεία προς τα και ζητήσαμε από την νομική υπηρεσία να μας υποβάλει την ε, γνωμοδότησή τη, πράγμα το οποίο θα κάνει τώρα. Uh, thank you, Mr. Sorry, you've been uh, described as the lady in the blue, but please, I'm sorry, I didn't have your name today. Uh, εσείς είστε, συγγνώμη, δεν είχα το όνομά σας. Hm? Να παρακαλώ, έχετε το λόγο. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε, αξιότιμοι κύριε Ευρωβουλευτέ. Όπω αναφέρατε, η Επιτροπή σα συζήτησε νομική γνωμοδότηση σε σχέση με την κοινή πορεία εμπρό για τα μεταναστευτικά θέματα ανάμεσα στο Αφγανιστάν και την Ευρωπαϊκή Ένωση. Το ερώτημα που τέθηκε στην νομική υπηρεσία αφορούσε τα εξή θέματα. Πρώτον, μπορεί αυτό το έγγραφο να θεωρηθεί ως διεθνή συμφωνία, όπως αναφέρεται στο τμήμα 5. Δεύτερον, τι επιπτώσεις έχει αυτό όσο κοινή πορεία μπροστά ε, και ε, μέτρα, οι δράσει ε, των θεσμικών οργάνων της Ένωση, των Οργανισμών ή των κρατών μελών επί τη βάση αυτού του εγγράφου έχουν παρόμοιε επιπτώσεις όπως αυτές της Συμφωνίας Επανεισδοχή και αν ναι, ποιες είναι οι πιθανές νομικές ε, λύσεις που μπορούν να δοθούν. Και τώρα, αν δεν θεωρείται διεθνή ε, συμφωνία αυτή η κοινή πορεία μπρος, ποιες είναι οι αρμοδιότητες του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Όπως αναφέρθηκε πριν, η νομική υπηρεσία ε, σας έστειλε την γνωμοδότησή της στις 17 Μαρτίου. Ας επανέλθω τώρα στο κοινή πορεία μπροστά. Εγκρίθηκε στις 2 Οκτωβρίου του 2016 από την Ευρωπαϊκή Ένωση και την Ισλαμική Δημοκρατία του Αφγανιστάν με υποτιμορφή τη μορφή διακήρυξης που αντικοτόπτριζε την κοινή δέσμευση και παραθέτω για εντατικοποίηση της συνεργασίας για την αντιμετώπιση και πρόληψη της παράνομης μετανάστευσης και σχέση με την επιστροφή των παράνομων μεταναστών. Για το θέμα του κατά πόσο η κοινή πορεία μπροστά μπορεί να θεωρηθεί ή όχι ως διεθνή συμφωνία, έχουμε εξετάσει αυτό το μέσο υπό το φως της νομολογίας του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου. Σύμφωνα με αυτή την νομολογία, το καθοριστικό κριτήριο για να ορίσουμε κατά πόσο αυτό το κείμενο είναι δεσμευτικό ή όχι, είναι η πρόθεση των μερών. Με άλλα λόγια, δεσμευτική επίπτωση μιας συμφωνίας βασικά εξαρτάται από την πρόθεση των μερών να δεσμευθούν από αυτό ή όχι, από αυτήν ή όχι, ως θέμα διεθνής, ως, μάλλον ε, να είναι διεθνής νομοθεσία. Επί τη βάση των όρων αυτής της συμφωνίας εξαρτά, ε, μάλλον ε, βασίζεται αυτή η δέσμευση και ε, σε σχέση με το πλαίσιο υπό το οποίο συντάχθηκε. Γιατί η κοινή πορεία εμπρό, η πρόθεση των μερών σαφώ εκφράζεται στους, ε, στο διδακτικό αυτού του εγγράφου που λέει ότι στόχο δεν έχει να δημιουργήσει νομικά υποχρεώσεις ή οι δικαιώματα υπό υποχρεώσει ή δικαιώματα υπό τη διεθνή νομοθεσία επιπλέον η δικαιωματα υπο τη διεθνη νομοθεσια επιπλεον η γλωσσα στην οποία συντάχθηκε αντικατοπτρίζει πρόθεση των μερών να υπογράψουν μια κοινή δήλωση και όχι ε, μια διεθνή συμφωνία. και αυτό επικυρώνεται υπό τις περιστάσεις υπό τις οποίες συντάχθηκε αυτό το έγγραφο. Υπογράφηκε από εκπροσώπους του διπλωματικού επίπεδου της κυβέρνησης του Αφγανιστάν και της Ευρωπαϊκής Αντιπροσωπείας του Αφγανιστάν. Είναι επίσης σημαντικό να αναφέρουμε ότι στις διεθνείς σχέσεις πρόκειται για πολιτική επιλογή της Ένωσης είτε να δεσμευθεί για, σε μια νομικώς δεσμευτική συμφωνία είτε να υιοθετήσει μια πολιτική δέσμευση. Και το ίδιο ισχύει και για το άλλο συμβαλόμενο μέρος. Δηλαδή, η τρίτη χώρα μπορεί να θέλει να προβεί σε δεσμευτική συμφωνία με την Ένωση ή μπορεί να προτιμά να συνεργαστεί με την Ένωση, αλλά επί τη βάση ενός μη δεσμευτικού πλαισίου. Ως αποτέλεσμα καταλήξαμε ότι η κοινή πορεία εμπρός εμπίπτει στην κατηγορία μέσων απαλής νομοθεσίας για συντονισμένες δράσεις. Αυτό ευρέως χρησιμοποιείται, τέτοιου είδους μέσα χρησιμοποιούνται στις διεθνείς σχέσεις και αυτού του είδους οι συμφωνίες επιτρέπουν στα ενδιαφερόμενα μέρη να εκφράσουν πολιτική ε, δέσμευση, αλλά χωρίς να προβούν σε νομικό δεσμευτική συμφωνία. Αυτά τα μέσα έχουν αναγνωριστεί και στην ομολογία του ε, δικαστήριου και μπορούμε να αναφέρουμε πρόσφατη απόφαση του του ε, δικαστηρίου σε σχέση με την δήλωση Ευρωπαϊκής Ένωσης Τουρκίας. Τώρα όσον αφορά τις επιπτώσεις αυτή τη δήλωση η Ευρωπαϊκή Ένωση και το Αφγανιστάν δεν είναι υποχρεωμένα να ακολουθήσουν τους όρου συνεργασία που ορίζονται σε αυτό έγγραφο. διαφορά σε σχέση με τις συμφωνίες επανεισδοχή. Αυτό, η κοινή πορεία εμπρό μπορεί να έχει πρακτικές επιπτώσεις όσον αφορά τη διευκόλυνση επανεισδοχής ε, Αφγανών που παρανόμως διαμένουν στην Ένωση. Αυτές οι επιπτώσεις μπορεί να είναι παρόμοιες με αυτές τις συμφωνίες επανεισδοχής, μόνο όμως με υπό τον όρο ότι τόσο η Ένωση όσο και το Αφγανιστάν σέβονται τους όρους συνεργασίας που ορίζονται ε, σε αυτό το έγγραφο κοινή πορεία εμπρό. Επειδή όμως αυτό το έγγραφο βασίζεται μόνο σε πολιτική ε, δέσμευση υπάρχει λιγότερη ε, βεβαιότητα από ότι στη Συμφωνία Επανεισδοχής και ότι δηλαδή θα γίνουν σεβαστοί οι όροι αυτοί. Τώρα, ε, ποιες μπορεί να είναι οι νομικές διορθώσεις. μπορούν τα ενδιαφερόμενα άτομα με βάση το άρθρο 13 της Οδηγίας περί επιστροφής ή σύμφωνα με την εθνική τους νομοθεσία να προσβάλλουν την απόφαση που θα ληφθεί επί τη βάση αυτού της κοινή πορεία εμπρό. Μια απόφαση επιστροφή προς το Αφγανιστάν θα πρέπει να λαμβάνει υπόψη, να εξετάζει μάλλον ξεχωριστά την κάθε υπόθεση και επίσης την κατάσταση που επικρατεί στη χώρα επιστροφής. Ακόμα και αν ληφθεί απόφαση περί επιστροφής αλλά υπάρχουν βάσιμοι λόγοι ώστε να πιστεύουμε ότι η επιστροφή των μεταναστών σε συγκεκριμένη χώρα, δηλαδή εδώ το Αφγανιστάν, θα παραβίαζε ε, την αρχή του non-refoulement, μια τέτοια επιστροφή λοιπόν θα πρέπει να ανασταλεί, να μην ε, υλοποιηθεί. Είναι σημαντικό λοιπόν ότι δεν είναι δεσμευτική, να πούμε ότι δεν είναι δεσμευτική αυτή η κοινή πορεία εμπρό και το σχετικό έγγραφο και δεν επηρεάζει την μεταναστευτική πολιτική της Ένωσης ούτε δημιουργεί νέε υποχρεώσεις. Σε σχέση με το θέμα των αρμοδιοτήτων του Κοινοβουλίου, η διαδικασία που προβλέπεται στο άρθρο 218 της συνθήκης δεν ισχύει, διότι η κοινή πορεία δεν αποτελεί διεθνή συμφωνία. Ωστόσο το Κοινοβούλιο φυσικά μπορεί να χρησιμοποιήσει τις δημοδιότητες που έχει ώστε να προβεί σε πολιτικές ενέργειες και όχι νομικές ενέργειες αν διαφωνεί με την πολιτική της Κομισιόν της σύναψης μέσων απαλής νομοθεσίας με τρίτες χώρες. Σας ευχαριστώ πολύ για την προσοχή σας και βεβαίως είμαστε στη διάθεσή σας για οποιαδήποτε ερώτηση μπορεί να έχετε. Μάλιστα, ευχαριστώ. Αυτό είναι ένα παράδειγμα για πράγματα που είναι τόσο σημαντικά να καταλάβουμε αλλά που είναι δύσκολο να τα καταλάβει κανείς. Τα προνόμια του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου είναι ζωτική σημασία εδώ και το σημαντικό είναι αυτό που λέτε στο τέλος. Σίγουρα όμως και πολλά άλλα είναι πολύ σημαντικά. Δεν θυμάμαι τώρα ποιο ήταν που είχε ζητήσει την γνωμοδότησή σας. Ε, Μπάρμπαρα, θες το λόγο, ξέρω ποιος άλλος. Η Μπάρμπαρα είναι η πρώτη και μετά η Σεσίλ. Ευχαριστώ Πρόεδρε και ευχαριστώ την νομική υπηρεσία για την νομική γνωμοδότηση που αποσαφηνίζει πολλά ε, ζητήματα κυρίως ε, σε σχέση με τι τι νομικές ε, διορθώσεις ή λύσεις μπορεί να υπάρχουν. Τώρα, αυτό που θέλω να ρωτήσω εγώ την νομική υπηρεσία είναι τα κίνητρα, τους λόγους μάλλον, για τους οποίους δεν έγινε μια ε, κλασική ε, διεθνή συμφωνία και επελέγει αυτή η προσέγγιση της του ατελούς ε, δικαίου. Είναι κάτι το οποίο μας ενδιαφέρει πολύ. Γιατί δεν επελέγει λοιπόν μια τέτοια συμφωνία. Είναι μια συμφωνία ε, Και αυτό οφείλεται στο ότι μέσα στην ευγανική κυβέρνηση επικρατούσαν βαθιές ε, αντιθέσεις όσον αφορά τη φύση αυτής της συμφωνίας. Ε, ε, μάλιστα αντιπαραθέσεις που ήταν πολύ έντονες και από ό,τι φαίνεται είχαν προβλεφθεί μαζικοί επαναπατρισμοί και μάλιστα ένα έγγραφο της, ε, της Υπηρεσίας ε, Εξωτερικής Δράσης μιλούσε για την επαναπατρισμό 80.000 Αφγανών ε, για μια οπότε η Σύμβαση της Γενέβης ε, ορίζει, που ορίζει με μονομένη εξέταση κάθε υπόθεση, κάθε περίπτωση ε, ασύλου ε, δεν τηρούνταν και η κυβέρνηση του Αφγανιστάν, ο υπουργό Εξωτερικών και ο υπουργό Μετανάστευση ήταν κατά των αναγκαστικών επιστροφών που προβλέπονται όμως από αυτό το joint way forward, την κοινή πορεία μπρο. Οι αναγκαστικές, αναγκαστικοί επαναπατρισμοί προβλέπονται ακόμα και για συνόδευτου ανήλικους Όλα αυτά λοιπόν βρίσκονται λίγο στα όρια της νομιμότητας. Και αυτά βρίσκονται, είναι μάλλον τα βασικά αίτια του ότι τέτοιου είδους συμφωνίες τελικά μεταφράζονται και μετατρέπονται σε ατελές δίκαιο, soft law, γιατί δεν μπορούν έτσι να ελεγχθούν ούτε από το Ευρωκοινοβούλιο, αλλά ούτε και από την τρίτη χώρα. και η νημική γνωμοδότηση λέει ότι το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο έχει τη δυνατότητα να αντισταθεί και να αντιπαρατεθεί, να θέσει ερωτήσεις, πράγμα που με χαροποιεί, αλλά κατά τη γνώμη μου δεν αρκούν οι ερωτήσεις, το έχουμε ήδη κάνει αυτό. Ε, και επισήμως. Γίνεται λόγος για τη σύσταση Επιτροπής Ερευνητικής. Εγώ και στο όνομα της ομάδας μου ζητώ να ξεκινήσει μια τέτοια, να συσταθεί μάλλον μια Επιτροπή Ερευνητική για αυτή την υπόθεση αυτή της συμφωνία που περιλαμβάνει ένα σωρό σημεία που περιλαμβάνει πολλά στοιχεία πολύ αμφισβητήσιμα σε σχέση με το διεθνές, δικαίωμα, ε, το διεθνές δίκαιο, όπως ας πούμε η μαζική επαναπατρισμού, παραβίαση της αρχής του non-refoulement και καταναγκαστικές επιστροφές επαναπατρισμοί. Όχι εθελοντική. Ευχαριστώ, Μπάρμπαρα. Είσαι σύλλο. Ευχαριστώ. Εγώ Είχαμε στην αρχή τη δήλωση Ένωση τη Τουρκία. Μετά έχουμε την κοινή πορεία εμπρό Αφγανιστάν Ένωση. Μέσα από αυτέ τι συμφωνίε ε, προχωρούμε στο όριο τη ε, δημοκρατική και η Κομισιόν ε, στην ουσία. Ε, ισορροπία ανάμεσα σε νομιμότητα και μη νομιμότητα. Ε, θα πρέπει δηλαδή να θεωρήσουμε πως αυτή η, κοινή αυτή η δράση το... με το Αφγανιστάν θα θεωρηθεί ως μια απαρχή για νέο είδους ε, τέτοιες δράσεις με άλλες υπο... Ε, ασφαλείς χώρες. Τώρα για τις εκατοντάδες, χιλιά... εκατοντάδες ε, συνόδευτους ανήλικους από το Αφγανιστάν για τους οποίους μίλησε πριν η συνάδελφος Βάρβαρα, να θυμίσω ότι έχουμε ένα σωρό ασυνόδευτους ανηλίκους στην Ιταλία που μάλιστα βρίσκονται στην περιφέρεια Φρίουλη Βενέτσια Τζούλια τι θα γίνουν εκεί πέρα, τι θα γίνουν αυτοί, προβλέπεται η επιστροφή τους, με ποιο τρόπο θα διευκολυνθεί η επιστροφή τους στην πατρίδα τους και θα ήθελα να γνωρίζω ακριβώς ε, αυτά τα ζητήματα πώς θα λυθούν με αυτή τη συμφωνία που δεν είναι συμφωνία. Ευχαριστούμε, Ιάννα. Ευχαριστώ. Όλα αυτά επιβεβαιώνουν αυτά που υποψιαζόμασταν. Ότι δηλαδή δεν νομιμοποιεί η συμφωνία αυτή κάτι που δεν θα μπορούσε να νομιμοποιηθεί. Δηλαδή καταναγκαστική επιστροφή ανθρώπων στο Αφγανιστάν που προφανώς δεν μπορεί να θεωρηθεί ασφαλής χώρα και προφανώς δεν ε, μπορεί να περιλαμβάνει ασφαλείς περιοχές. Συνεπώς, ήμουνα ένας, μία από τους βουλευτές που είχαν συνυπογράψει την προφορική ερώτηση και συμφωνώ με αυτά που είπε η Μπάρμπαρα, ότι δηλαδή όντως χρειαζόμαστε μια εξεταστική επιτροπή η Κομισιόν και το Συμβούλιο πρέπει να απαντήσουν για συγκεκριμένες περιπτώσεις που έχουν υλοποιηθεί, επιστροφές δηλαδή που έχουν υλοποιηθεί. Και ποιες είναι οι επιπτώσεις της πρακτικής αυτής που ακολουθείτε βάσει αυτή της μη δεσμευτικής συμφωνίας που υπογράφηκε με πρόθεση να κορυδέψει τελικά την ευρωπαϊκή κοινή γνώμη ότι δηλαδή υπάρχει μια συμφωνία για μασικές επιστροφές. Είναι ασύμβατο αυτό με το διεθνές δίκαιο. Είναι ασύμβατη αυτή η συμφωνία με τις υποχρεώσεις των χωρών μελών μας. Και θέλω να ξέρω τι έγινε με τις συγκεκριμένε περιπτώσεις, με τους ανθρώπους αυτούς που επιστράφηκαν δηλαδή στο Αφγανιστάν. Και πώς ε, μπορούμε να διορθώσουμε το κακό. Οι χώρες μέλη που επέτρεψαν στους αυτούς τους να προβούν στις επιστροφές αυτές λογοδοτούν. Ιδιαίτερα αυτό που με απασχολεί είναι ότι πολλές από τις περιπτώσεις των ανθρώπων που φεύγουν από το Αφγανιστάν και προσπαθούν να βρουν μια νέα ζωή στην Ευρώπη είναι άνθρωποι που συνεργάστηκαν, κάποιοι τουλάχιστον από αυτούς, με την Διεθνή Συμμαχία στο Αφγανιστάν. Ήταν διερμηνείς των στρατευμάτων εκεί είναι άνθρωποι οι οποίοι είναι πάρα πολύ ευάλωτοι. Κινδυνεύουν. Γιατί επειδή ήταν διερμηνείς, υπηρέτησαν δίπλα ε, στις ε, δυνάμεις των συμμάχων και επιτόπου δεν τους προστατεύουν. Οπότε προφανώς και δεν πρέπει τέτοιοι άνθρωποι να επιστρέφονται στο Αφγανιστάν που είναι μια χώρα που δεν είναι ασφαλής. Ευχαριστούμε. Ευχαριστώ. Θέλω να επενθυμίσω κάποια πράγματα όσον αφορά την συμφωνία με την Τουρκία. Ε, θα έπρεπε να έχει και εκεί συμμετέχει το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Τι κάνανε, μας πήραν μαζί. Όχι. Σταμάτησαν να μιλάνε για αυτή τη συμφωνία και άρχισαν να τη λένε δήλωση. Δεν θα είμαστε ικανοποιημένοι με αυτό το μοντέλο με το Αφγανιστάν, με τη Λιβύη, με άλλες αφρικανικές χρόνες, όπου κάθε φορά λέγεται ε, ένα άλλο πλαίσιο όπως το, αυτό το σύμφωνο για την μετανάστευση. Αυτό που κάνουμε τι είναι, ε, αναθέτουμε σε άλλους τη φροντίδα των συνόρων μας και αναθέτουμε σε άλλους τις ευθύνες μας. Αντίθετα με τις δεσμεύσεις που αναλάβαμε πέρσι στην Νέα Υόρκη για μεγαλύτερη και καλύτερη κατανομή των ευθυνών για την υποδοχή για το άσυλο, ενώ το γεγονότο το 86% των προσφύγων αυτή τη στιγμή φιλοξενούνται στις πιο φτωχές περιοχές του κόσμου. Στην ουσία θυσιάζουμε με αυτόν τον τρόπο και για αυτούς τους λόγους τις σχέσεις μας με, τα τρίτε με τις τρίτες χώρες. Ε, θυσιάζουμε και τις αρχές μας ε, που είναι γεγραμμένες στο χάρτη θεμελιωδών δικαιωμάτων. Εμείς ε, θυσιάζουμε την ουσία της αναπτυξιακής πολιτικής της Ευρωπαϊκής Ένωσης που ο βασικός στόχο έχει να εκριζώσει τη φτώχεια, όχι να διαχειριστεί και να ελέγξει τα σύνορα. Εμείς στην Επιτροπή Ανάπτυξης, συνάδελφοι, ε, φτιάξαμε μια ομάδα εργασίας που είναι ειδικά φτιαγμένη για να δει πώς με βάση αυτές τις συμφωνίες τα κονδύλια για την ανάπτυξη χρησιμοποιούνται για στόχους διαχείρισης συνόρων και για την οικοδόμηση δυνατοτήτων. Είμαι πολύ ικανοποιημένη που η γνωμοδότηση αυτή νομική θυμίζει πως το Κοινοβούλιο, αν και δεν ε, ε, συμμετέχει άμεσα μπορεί να χρησιμοποιήσει άλλα μέσα, δηλαδή μπορεί να ασκήσει έλεγχο στον προπολογισμό. Και εδώ περιοριζόμαστε όμως λόγω τη περιπλοκότητας και της αδιαφάνειας αυτών των νέων μέσων χρηματοδότηση, όπως εκείνα τα καταπιστέματα ή το νέο σχέδιο επενδύσεων για την Αφρική. Σας καλώ όλους να μα στηρίξετε στη δουλειά που κάνουμε στην Αναπτυξιακή Επιτροπή για το πώ χρησιμοποιούνται αυτά τα κονδύλια και γιατί είδου project, ώστε να αφιερώνονται πραγματικά πραγματικά στην κρίση της φτώχειας και όχι για να δημιουργούν και άλλους τείχους που αυξάνουν την φτώχεια. Ευχαριστούμε πολύ, Ευχαριστώ την νομική υπηρεσία για την γνωμοδότησή της. Υπογραμμίζει αυτά τα οποία έτσι καλώς γνωρίζαμε και που τόσο εύλογα τα είπε και η Μπάρμπαρα και τον Σικέλη Τι περιλαμβάνει αλλά το θέμα είναι, όπως είπε και η Μπάρμπαρα, ότι μας αφαιρούνται τα προνόμια μας. Συνεπώς το στοιχείο κλειδί εδώ, και συγγνώμη, έπρεπε να το είχα πει και στην αρχή, Το θέμα των προνομίων μας είναι ζωτική σημασία και γι' αυτό έχουν συμμετάσχει όλα τα μέλη και εξετάζουμε την στρατηγική, τη ρεαλιστική στρατηγική μπορούμε να έχουμε, γιατί όλοι είσαστε ρεαλιστές. Κάποια πράγματα δεν μπορούμε να κάνουμε, μπορούμε να φωνάζουμε, αλλά πρέπει να έχουμε μια στρατηγική και η Έλλη έδωσε μια ιδέα. Λοιπόν, το πρώτο που θέλω να πω είναι και είναι σημαντικό να διασφαλίσουμε ότι οι άνθρωποι εδώ, οι πολιτικοί γνωρίζουν ότι μας έχουν αφαιρεθεί προνόμια. Και μετά χρειαζόμαστε μια στρατηγική. Αλλά προτιμώ η στρατηγική αυτή να γίνει με αυτούς οι οποίοι έχουν ασχοληθεί με το θέμα, έτσι ώστε η στρατηγική μας να είναι καλά επικεντρωμένη. Να μην την να μην αφήσουμε τα πράγματα στα χέρια του Συμβουλίου και της Επιτροπής. Έχει να κάνει με τις πολιτικές μας, ναι, αλλά έχει να κάνει με τα προνόμια μας. Σας ευχαριστώ για αυτή τη συζήτηση. Στους συντονιστέ. θα το συζητήσω, θα το ζητήσω μια στρατηγική. Πώς θα αποφύγουμε τέτοιου είδους μοντέλα τελούς δικαίου που μας αφαιρούν τα δικά μας δικαιώματα, τα δικά μας προνόμια. Λοιπόν, ευχαριστώ πολύ. Τώρα δεν ξέρω αν η Επιτροπή... Νομίζω ότι είναι καλύτερα να προχωρήσουμε γρήγορα, να πάμε στην επόμενη συνάντηση των συντονιστών και να το βάλουμε εκεί το θέμα. Να αξιολογήσουμε δηλαδή το τι κάνουμε από εδώ και πέρα γιατί θέλω γρήγορα η ομάδα επαφή για το άσυλο να αντιδράσει. Δεν θέλω να μπαίνει στην ημερήσια διάταξη ξανά και ξανά και να μην έχουμε στρατηγική. Ωραία, σας ευχαριστώ πολύ λοιπόν. Ευχαριστώ και την νομική υπηρεσία κύριε Παντός και σας ευχαριστώ πολύ. Και φτάνουμε στο σημείο 5 Πρόκειται για την αξιολόγηση του REFIT όσον αφορά το νομικό πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Χαίρομαι που είσαστε εδώ ακόμα υπομονετικά. Λοιπόν, πρόκειται για την αξιολόγηση ρέφητο, όπω είπαμε, όσον αφορά το νομικό πλαίσιο τη Ευρωπαϊκή Ένωση κατά τη υποβοήθηση τη παράνομη εισόδου, διέλευση και διαμονή δέσμη μέτρων για τους διακινητές παρανόμων μεταναστών και είναι η οδηγία 2290 και απόφαση πλαίσιο 2002-946 ακριβώς για την υποβοήθηση αυτή τους διακινητές ε, παράνομων μεταναστών κλπ. Εδώ λαμβάνουμε υπόψη τη εξελίξη τι έχει γίνει με το πακέτο ε, διευκόλυνσης και θα δώσω το λόγο. Στην κυρία Τυράτση από την DG Home που θα μας παρουσιάσει την αξιολόγηση αυτή, κυρία Τσιράτσι. Παρακαλώ και συγγνώμη που αργήσαμε. Θέλουμε να μας δώσετε, να μας συνοψίσετε, κύριε Τσινάτση. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Όπως είπατε και εσείς, στόχος της αξιολόγησης αυτής είναι να δούμε δύο εργαλεία που έχουμε στη διάθεσή μας πώς λειτουργήσαν. Δηλαδή η οδηγία 90 και η απόφαση πλαίσιο 946. Αν ανταποκρίνονται στους στόχους μας. Χρησιμοποίησαμε διάφορα κριτήρια για να μετρήσουμε την αποτελεσματικότητα, τη συνοχή και την προσθέμενη αξία που προσφέρουν αυτά τα εργαλεία. Θα αναφερθώ πρώτα στην μεθοδολογία για να δούμε πώς φτάσαμε στα συμπεράσματα στο οποία φτάσαμε. Ε, πρόκειται για μια αξιολόγηση που έγινε το 2015 και 2016 και στηρίχτηκε από μια ε, έκθεση και αξιολόγηση που είχε γίνει σε διεθνή φόρα, διεθνείς οργανώσεις, από την ίδια την Ευρωπαϊκή Επιτροπή νωρίτερα σε άλλες αξιολογήσεις που είχαμε κάνει. Επίσης, χρησιμοποίησαμε και δύο εξωτερικές μελέτες για να δούμε ποια είναι τα χαρακτηριστικά της ε, ενσωμάτωσης στο εθνικό δίκαιο. Πώς έγινε αυτή η ενσωμάτωση. Επίσης, είχαμε και ανοιχτή διαβούλευση, στοχευμένη, διαβούλευση με τις χώρες μέλη, τις αρχές των χωρών μελών, με διεθνείς οργανώσεις, μη κυβερνητικέ οργανώσεις, όπως επίσης και ανοιχτή με το κοινό διαβούλευση. Οι μελέτες στις οποίες ε, βασιστήκαμε εξέτασαν την αποτελεσματικότητα της ενσωμάτωσης στην εθνική νομοθεσία. Οι δύο μελέτες στις οποίες βασιστήκαμε είναι έτσι κι αλλιώς ανοιχτές στο κοινό και υπάρχουν στην ιστοσελίδα της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, οπότε μπορείτε να τις συμβουλευτείτε πλήρως με τα συμπεράσματα, με τα δεδομένα τα οποία χρησιμοποιήθηκαν, τα εμπειρικά και άλλα. Τώρα, δύο λόγια στη βάση που χρησιμοποιήθηκε για την μελέτη, γιατί είναι σημαντικό να ξέρουμε πώς φτάσαμε στα συμπεράσματά μας. Τα δεδομένα που χρησιμοποίησαμε ήρθαν από τη Frontex, την Eurostat ε, και άλλες έρευνες που έχουν γίνει. Ερωτηματολόγια στάλησαν σε όλες τις χώρες μέλη. Τη συζητήσαμε με οργανώσεις του ΟΗΕ, με την Europol, ε, με μη κυβερνητικέ οργανώσεις ε, στην Ισπανία και αλλού. Συζητήσαμε επίσης με εκπροσώπους και διεθνών οργανισμών και επιχειρήσεων και είχαμε και τέσσερις συγκεκριμένες περιπτώσεις ε, που αναλύσαμε πιο συγκεκριμένα. Οργανώσαμε επίσης ως Επιτροπή συναντήσεις υπό τη μορφή διάφορων φόρα με διάφορες πλευρές. Πάντα στόχος μας ήταν να διασφαλίσουμε ότι βασιζόμαστε σε όσο γίνεται ευρύτερο φάσμα πληροφοριών. Είναι ένα θέμα που έτσι καλλιώς ε, τα τελευταία χρόνια συζητήθηκε πολύ. Οπότε και το κοινό έχει δείξει ενδιαφέρον, γι' αυτό θέλουμε και τις απόψεις του κοινού. Είχαμε λοιπόν, όπως σας είπα, ερωτηματολόγιο, στο οποίο συμπεριλαμβάναμε το θέμα της ε, λαθροδιακίνησης πήραμε 2.425 απαντήσεις και πάνω από το 95% ήταν ιδιώτες που απάντησαν. Κάτι το οποίο δείχνει πόσο μεγάλο ενδιαφέρον δείχνει ο κόσμος, οι πολίτες μας σε αυτό το συγκεκριμένο θέμα. Ποια ήταν τα συμπεράσματα τώρα της αξιολόγησης. Πρώτον, ένα το οποίο ε, θα πρέπει να μας δάξει πολλά είναι αυταπόδεκτο. Δηλαδή, από τις μελέτες που έγιναν, από τις διαβουλεύσεις που κάναμε, φάνηκε ότι υπάρχει μια δυναμία όσον αφορά τα δεδομένα, τη συλλογή δεδομένων δηλαδή που έχουν διάφορες αρχές. Και αυτό πρέπει να διορθωθεί αν θέλουμε οι αποφάσεις μας να βασίζονται σε πλήρη στοιχεία. Το δεύτερο συμπέρασμά μας ήταν το θέμα των κυρώσεων όσον αφορά την κακή ενσωμάτωση της νομοθεσίας. Οι κυρώσεις αυτές δεν ήταν αποτελεσματικές, γιατί όσον αφορά την αποτελεσματικότητα εμείς ε, διαπιστώσαμε ότι δεν επηρέασε η ενσωμάτωση αυτή, στην καλύτερη των περιπτώσεων ήταν ουδέτερη. Όσον αφορά τώρα τον ορισμό της παράβασης αυτής της λαθροδιακίνησης. Εδώ υπήρχαν επικρίσεις για την έλλειψη νομικής βεβαιότητας όσον αφορά την ανθρωπιστική βοήθεια και την ε, διευκόλυνση. Μη κυβερνητικέ οργανώσει. αντιμετώπισαν δυσκολίε κάποιε από αυτέ στη Μεσόγειο που προσπάθησαν να διασώσουν ε, μετανάστες. Το θέμα της ανθρωπιστική αρρωγής τώρα. Αυτό που κάνει ο Διγέν ότι προσφέρει την επιλογή όσον αφορά την ε, είσοδο ανθρώπων και την ε, βοήθεια που τους προσφέρεται. Για 7 χώρες υπάρχουν κάποιες εξαιρέσεις στην νομοθεσία και ανάμεσα σε αυτές τις 7 χώρες όλες είναι στην πρώτη γραμμή και υποδέχονται στη Μεσόγειο Ιταλία, ε, Μάλτα, Ελλάδα, Ισπανία και κάποιες άλλες χώρες μέλη. Πρέπει επίσης να έχουμε υπόψη μας ότι η βοήθεια στους έχοντες ανάγκη είναι μια υποχρέωση. Δεν είναι κάτι που εξαρτάται από το πώς θα εφαρμόσει κανείς την νομοθεσία. Δεν τίθεται θέμα δηλαδή πώς ε, θα ερμηνεύσει, θα εφαρμόσει κτλ. Όσον αφορά λοιπόν τις μη κυβερνητικές οργανώσεις που βοήθησαν στη διάσωση ε, ανθρώπων στη θάλασσα, έχουν την υποχρέωση να το κάνουν. Μα απασχόλησε αποτελεσματικότητα, όπω είπαμε και στην αρχή. Επειδή όμω δεν υπάρχουν ε, πάντα σωστά δεδομένα, ήταν δύσκολο να καταλήξουμε σε ένα συμπέρασμα. Αυτό όμω που φάνηκε σαφώ είναι ότι το κόστος της λαθροδιακίνησης είναι τεράστιο, κάτι το οποίο απαιτεί νομική αντιμετώπιση από πλευράς Ευρωπαϊκής Ένωσης. Και όσον αφορά την προσθέμενη αξία της Ευρώπης, αυτό υπογραμμίστηκε από όλους όσοι απάντησαν. Είναι πολύ σημαντικό, όλοι λένε ότι χρειάζεται ένα πλαίσιο συνεργασίας σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης και για τις παρεμβάσεις και για τα μέτρα που λαμβάνονται. Για τη συνοχή ήταν θετική η απάντηση που είχαμε, η ουδέτερη. Και υπήρξε το θέμα της ε, συμπληρωματικότητας της οδηγίας με άλλα μέσα που διαθέτει η Ευρωπαϊκή Ένωση. Το συμπέρασμα λοιπόν της αξιολόγησης και το συμπέρασμα στο οποίο καταλήξαμε και εμείς και ο Επίτροπος Αβραμόπουλος όταν ήρθε εδώ αναφέρθηκε σε αυτό το Μάρτιο ήταν ότι η νομική αναθεώρηση δεν θα αποτελέσει προστιθέμενη αξία. Περισσότερη σημασία έχει η σωστή εφαρμογή των όσων ήδη έχουμε στη διάθεσή μας εδώ και δύο χρόνια. Και θα θέλαμε αυτόν να υπογραμμίσουμε. Τέλος, για τα επόμενα βήματα και για το πώς εμείς βλέπουμε τα επόμενα βήματα μετά από την αξιολόγηση αυτή. Να καλυφθούν οι δυναμίες όσον αφορά τα δεδομένα. Το συστάμε και με τη Eurostat για τα δεδομένα του 2017 και τώρα αρχίζουμε να παίρνουμε κάποια στοιχεία και είναι ένα πολύ σημαντικό βήμα γιατί τα σωστά στοιχεία μας επιτρέπουν να καταλήξουμε και σε πιο σωστές αποφάσεις. Η συνεργασία επίσης με τις χώρες μέλη και τις διάφορες οργανώσεις είναι κάτι που βοηθάει να βελτιωθούν τα δεδομένα που στηρίζουν τις πολιτικές μας. Η άλλη κατηγορία βημάτων για το μέλλον είναι η ανθρωπιστική αρρωγή. Ακόμα και αν το συμπέρασμα είναι ότι δεν θα πρέπει να αλλάξει η οδηγία που αναφέρεται στην ανθρωπιστική οδηγία, παρόλα αυτά αυτό πρέπει να αλλάξει είναι ο τρόπος με τον οποίο εφαρμόζεται αυτό λοιπόν προσπαθούμε και εμείς να κάνουμε τώρα. Συνεργαζόμαστε με τις χώρες μέλη, με τη Eurojust, με τις οργανώσεις ανθρωπίνων δικαιωμάτων, την κοινωνία των πολιτών, ώστε να διασφαλίσουμε ότι η νομική βάση όντως εφαρμόζεται και δεν γίνονται καταχρήσεις. Και τέλος, πρόγραμμα δράσης για την καταπολέμηση της ηλεκτροδιακίνησης. Είναι πολύ σημαντικό έχει στόχο το 2020 και εμείς θα κοιτάξουμε πολύ προσεκτικά το πώς εφαρμόζεται. Ε, σας ευχαριστώ. Ε, πρόκειται να σας ερωτήσω για το βασικό θέμα, το θέμα που απασχολεί τα μέλη μας. Διώξεις μη κρατικών οργανώσεων που προσφέρουν ανθρωπιστική βοήθεια καμιά φορά. Ποιος θα ήθελε, να ρωτήσω, εάν στην αξιολόγηση αυτή που κάνετε έχετε λάβει υπόψη τις επιπτώσεις του να τροφοδοτούνται τα δίκτυα των διακινητών επειδή οι χώρες μέλη δεν διαθέτουν νόμιμες ελεγχόμενες οδούς για την διέλευση προσφύγων και μεταναστών. Σεσίλ, εσείς, κύριε Κένγκε. Εγώ ήθελα να εξηγήσω γιατί ε, αυτή τη φάση, κυρίως στην Ιταλία που πρωταγωνιστεί σε όλη αυτή την ε, τρελή υπόθεση, να σας πω τι συμβαίνει. Πριν από κάποιες με, από λίγες μέρες είχαμε και μία συνάντηση και κλεισμένων των θυρών με τον Γενικό Εισαγγελέα και μας εξήγησε στην Κατάνια τι ακριβώς συμβαίνει με τη ΜΚΟ έλεγε λοιπόν ότι η ΜΚΟ ε, κάνοντας αυτό, πηγαίνοντας κοντά στις ακτές, ε, σώζοντας κόσμο, στην ουσία τι έκανε, αυξάνονταν οι μετανάστες. Και άρα το γεγονό ότι είχαμε αύξηση των μεταναστών τις τελευταίες εβδομάδες θυμίζω ότι ξεπεράσαμε τις 7.000 σε λίγες μόλις μέρες. Την εβδομάδα του Πάσχα είχαμε 8.000 αποβάσεις. Ε, τώρα σε μια εβδομάδα ακόμα 7.000 κόσμος. Ε, και όλα αυτά ξεκινούν από το γεγονός ότι ε, υπήρχαν μέσα που φτάνανε και μέχρι τι ακτέ τη Λιβύη. Αυτή τη συζήτηση με κεκλεισμένο των θυρών, Λίγες μέρες μετά την είδαμε στις εφημερίδες σε πόνημα. Προς έκπληξή μας λοιπόν βρεθήκαμε ενώπιον μιας κοινή γνώμης, ε, δημοσιογράφοι, κοινωνία των πολιτών, πολλοί άρχισαν να τροφοδοτούν αυτή τη συζήτηση ότι αυτοί η ΜΚΙΟ, ότι οι ΜΚΙΟ μάλλον βοηθάνε τους ε, ε, διακινητές. Όμως αυτά πρέπει εμείς να τα διερευνήσουμε. Ποιες, ποιοι είναι οι κανόνες στις οποίες θα πρέπει να υπακούμε και να υπακούν αυτέ οι ΜΚΟ. Ξεκινώντα από το γεγονό ότι υπάρχει υποχρέωση διάσωση. Δεν μπορούν δηλαδή να κάνουν πώ δεν βλέπουν τον κόσμο που βρίσκεται εκεί. Ποιοι είναι οι κανόνε στου οποίου θα πρέπει να υπακούν οι ΜΚΟ για να λένε ότι λειτουργούν με πλήρη διαφάνεια. Γιατί ούτω ή άλλω είναι υποχρεωμένοι να σώσουν τον κόσμο που κινδυνεύει στη θάλασσα. Ο εισαγγελέα λοιπόν θα έπρεπε να μα δώσει τελικά το πόρισμα τη έρευνα και όχι να αναφέρει όλο αυτό το ερώτημα. Όταν ρωτήσαμε ποια είναι τα στοιχεία, μας είπε όχι, υπάρχουν υποψίες. Άρα λοιπόν το θέμα είναι άλλο. Τα κράτη-μέλη δεν έχουν πληρώσει πολιτικά από την κρίση της αλληλεγγύης αυτή το κενό που τώρα καλύπτουν η ΜΚΟ. Δεν μπορούμε λοιπόν να δαχτυλοδείχνουμε αυτούς που στην ουσία καλύπτουν τα κενά και περιμένουμε κανόνες. Αν θέλουμε πραγματικά να σώσουμε τον κόσμο, πρέπει πρώτα απ' όλα να είμαστε σαφεί. Όχι ότι οι ΜΚΟ βοηθάνε του διακινητέ. Ποιοι είναι οι κανόνε που πρέπει να τηρούν οι ΜΚΟ με τι αλλαγέ και με την κρίση που διανύουμε αυτή τη στιγμή όσον αφορά την κινητικότητα. Τι, τι, τι, κά, κά, κάποιοι πρέπει να είναι συγκεκριμένοι οι κανόνες στου οποίου θα πρέπει να υπακούν οι ΜΚΟ. Είναι τρελή αυτή η κατάσταση που ζούμε, κατά τη γνώμη μου, όπου οι ένοχοι είναι αυτοί οι οποίοι καλύπτουν ένα πολιτικό και νομικό κενό, το οποίο πρέπει γρήγορα να καλύψουμε. Ευχαριστώ. Σύντομα, να παρακαλώ. Ναι, εγώ ήθελα μετά από αυτά που είπε η Σίλια να πω για αυτούς που σκέφτονται ε, και ενοχοποιούν ΜΚΟ που σώζουν ζωές στη Μεσόγειο, μήπως προτείνουν να ενοχοποιηθούν και η θαλάσσια επιχείρηση της ε, CSDP που σώζει χιλιάδες κόσμο επίσης στη Μεσόγειο. Γιατί ναι, όσο πιο πολλές ζωές ε, σώζεις, Βέβαια, θα ρίνεις κι άλλους να διασχίσουν τη Μεσόγειο. Αν αυτή είναι η, η, τρελή λογική, είναι... Είναι πραγματικά παράλογα όλα αυτά τρελά, εξωπραγματικά, όπως είπε και η Σεσίλια. Όπως είπε και η κυρία Κέγκε, δεν καταλαβαίνουμε ποια είναι η νομική θέση που ενοχοποιεί τη ΜΚΟ. Αυτό δημιουργεί περισσότερη ε, πολιτικά και φιλοσοφικά προβλήματα. Εσείς μας είπατε που κατευθύνεται η Κομισιόν. I'm not sure where to take this now, but I think. Sorry, sorry. Could you please respond? I'm getting tired. It's a short. Α, συγγνώμη, συγγνώμη, αρχίζω να κουράζομαι. Μπορείτε να απαντήσετε σε όλα αυτά, τις παρατηρήσεις. Σας ευχαριστώ πολύ, Πρόεδρε. Με ρωτάτε να πω πού βρισκόμαστε. Ο τρόπος με τον οποίο εξελίσσεται η κατάσταση στην Ιταλία δεν έχει να κάνει με τον νομικό κόρισμο και την ανάπτυξη της οδηγίας. Πιστεύουμε πως ήταν απαραίτητο να ξανανοίξουμε αυτή την οδηγία. Πιστεύουμε ότι οι κανόνες για το πώς κανείς ε, θα πρέπει να ενεργήσει στη θάλασσα είναι σαφή. Δεν απορρέουν από την οδηγία εξάλλου, αλλά από διεθνείς νομικές υποχρεώσεις. Και η ΜΚΟ που ε, κάνουν σημαντική ανθρωπιστική δουλειά στην Μεσόγειο θα πρέπει να συνεχίσουν να την κάνουν. Παρομοίως, ε, η MED που αναφέρθηκε λειτουργεί με σαφείς κανόνες. Δεν υπάρχει κανένα πρόβλημα ή δυσκολία που να προκύπτει από την ε, έλλειψη κανόνων. Αυτό που είναι σημαντικό είναι ότι η συνεργασία των όσων προβαίνουν σε επιχείρηση τη διάσωση είναι ουσιαστική, είναι πολύ σημαντική, είτε πρόκειται για καπετάνιους εμπορικών πλοίων, για ΜΚΟ που λειτουργούν στην Μεσόγειο, είτε είναι η UNAFORMED, Όλοι πρέπει να, να συμμετέχουν στις συντονιστικές προσπάθειες που καταβάλλονται όπου έχουμε επενδύσει πολύ και εμεί ω Ένωση τα τελευταία δύο χρόνια, γιατί μόνο με αυτόν τον τρόπο μπορούμε να εξασφαλίσουμε ότι δεν θα υπάρχουν γκρίζε ζώνες όπου να μπορεί ο κανεί να τι ερμηνεύει όπω θέλει. Ταυτόχρονα θα πρέπει να πούμε ότι τίποτα ούτε στις οδηγίες ούτε στις εθνικές νομοθεσίες εμποδίζει τις, νομικές, ε, τις δικαστικές αρχές να ερευνήσουν για τις ιδιαιτερότητες ε, κάθε υπόθεσης. Ε, γι' αυτό μπορούν και να το κάνουν οι αρχές των κριτών μελών. Η οδηγία έτσι έχει τώρα ή αν ξαναδιατυπωθεί δεν τους εμποδίζει να κάνουν κάτι τέτοιο. Είναι εθνική αρμοδιότητα να διεξάγουν έρευνες επί τη βάση καταγγελιών. Και σε αυτό θα πρέπει οι δικαστικές αρχές της Ιταλίας να ε, εστιάσουν σε αυτές τις υποθέσεις που έχουν προκύψει εκεί. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ Σεσίλη. ευχαριστώ Άννα. Ολοκληρώνεται έτσι η μυρισία μας διάταξη. Διάφορα υπάρχουν. Όχι. Ωραία. Επόμενη συνεδρίαση προβλέπεται για την 11η Μαΐου. Τέλος της συνεδρίασης.